Colleagues, Καλώς ήρθατε στην δεύτερη μέρα της υποεπιτροπής μας ασφάλειας και άμυνας. Το πρώτο σημείο της σημερινής ημέρας διάταξης το εξετάζουμε από κοινού με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων Καλωσορίζουμε λοιπόν τον David Μακάλιστερ, τον πρόεδρο της ΑΦΕΤ και βεβαίως έχουμε και τους εκπροσώπους των αντιπροσωπιών για τις σχέσεις με την Βοσνία Ερζεγοβίνη και το Κόσοβο. Έχουμε ένα σημαντικό πάνελ για το Ελθία και την κατάσταση ε, στη Βοσνία Ζεγοβίνη πριν από την ε, αποστολή ad hoc στη Βοσνία που θα γίνει αμέσως μετά το Πάσχα. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον David Μακάλιστερ, τον πρόεδρο της ΑΦΕΤ. Ευχαριστώ, Άννα Φωτίγκα. Ε, θα σας ξαναδώσω πολύ γρήγορα το λόγο και εγώ να σας καλωσορίσω. Είναι πολύ καλό ότι εξετάζουμε το θέμα της ασφάλειας στη Βοσνία και Ζεγοβίνη ως πρώτο σημείο σήμερα. Μετά θα δούμε τη στρατηγική επικοινωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια γενικότερα. Είναι κάτι που θα βοηθήσει εν ώψη και της επίσκεψης ε, ε στην μεγαλύτερη και πιο παλιά αποστολή ε, εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, στη Βοσνία δηλαδή, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον έχει παρουσιάσει τη στρατηγική Δυτικά Βαλκάνια, έχει διάμεση αξιολόγηση για, το, την προταξιακή ενίσχυση και έχουμε και την έκθεση προόδου ε, για τη συνοδοκορφή τη Σόφια. οπότε καλό είναι να δούμε ε, και το, την κατάσταση στη Βοσνία προ προπίσμα τη ασφάλεια και τις ευρύτερε επιπτώσει που έχει αυτό. Ε, να προχωρήσουμε και να δώσουμε το λόγο στους ο ομιλητές μας θα έλεγα. Επιτρέψτε μου να καλωσορίσω ε, τα μέλη του πάνελ. Τρία μέλη έχουμε εδώ. Πρώτα ο κύριος Ζακ ε, Φχαντά, ε, προϊστάμενος στο τμήμα του Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδιασμού, ε, τον Γκέορκ Τσίγκλερ, αναπληρωτή προϊστάμενο της μονάδας ε, ε, για την Αλβανία και την Βοσνία Ζεγοβίνη στην Κυρία και τέλος βεβαίως ε, ο εκπρόσωπος ε, του ΝΑΤΟ, ο αντισυνταγματάρχης Νικολά Σαλό, ο οποίος είναι στρατιωτικός επίκουρος του υποδικητή της ανωτέρας συμμαχικής διοικήσεως. Λοιπόν, U4 Althea γενικά και η κατάσταση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στη Βοσνία Τζεγοβίνη. Πρώτα θα δώσω το λόγο στον Ζακ Φραντά Παρακαλώ. Καλημέρα σε όλους και όλες. Είμαι ο Ζακ Φραντά επικεφαλής της μονάδας στρατηγικής εξετάζουμε τις διαχειρίσεις κρίσεων στο πλαίσιο της CSDP e ε, και θα περιγράψω ε, ποιες είναι οι τάσεις αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την επιχείρηση Αλθέα. Θα σε ενημερώσω ε, για το θέμα αυτό, αλλά θα ήθελα πρώτα να το, να το θέσω σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Όπως ξέρετε, μετά από 10 χρόνια τα Δυτικά Βαλκάνια έχουν επιστρέψει στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κάνει μια προσπάθεια να επανεργοποιήσει τι μεταρρυθμίσει της χώρα των Δυτικών Βαλκανίων και να, ξανα, να ξαναμπούν στον δρόμο για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μήνυμα δόθηκε με, το, με την ομιλία του 2017 του, του κυρίου Γιούγκερ που μίλησε για την προοπτική την ανταξιακή των Δυτικών Βαλκανίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια στρατηγία για τα Δυτικά Βαλκάνια με ένα σαφέ δρόμο, ένα σαφές μονοπάτι για την ένταξη των χωρών αυτών, μεταξύ των οποίων και την Βοσνία Ερζεγοβίνη. Αυτή η στρατηγική είναι ένα μήνυμα προ την περιοχή για την βούληση τη Ευρωπαϊκή Ένωση να του δώσει μια αξιόπιστη προοπτική ένταξη. Η Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι μια μοναδική θέση από τι έξι αυτέ χώρε. Είναι η μόνη χώρα που έχει ε, στρατιωτική παρουσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση με συγκεκριμένη εντολή και Ηνωμένα Έθνη ε, για λόγου ασφαλείας για να αντιμετωπίζονται οι όποιε επιδεινώσεις της κατάσταση. Το ισχύει και για το Κόσοβο, αλλά αυτό είναι υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ. Σε ό,τι αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια τώρα και την Βοσνία Ζεγοβίνη, το Συμβούλιο ζήτησε μια αναθεώρηση στρατηγικής της επιχείρηση Αλθέα, λαμβάνοντα υπόψη ότι η Βοσνία Ζεγοβίνη έχει σημειώσει πρόοδο στην ενταξιακή ε, προσπάθειά τη και να υπόψη και την κατάσταση τη ασφάλεια στη χώρα. Όπως θα γνωρίζετε, η πρόοδος της επιχείρησης επανεξετάζεται κάθε έξι μήνες. Η στρατηγική αυτή αναθεώρηση που ε, κάναμε ήταν σε βάθος για πρώτη φορά ε, από τότε που υπάρχει επιχείρηση Αλθέρα το 2004 όταν έφυγε η δύναμη σταθεροποίηση του ΝΑΤΟ ε, για να βοηθήσουμε εμεί ε, τι αρχέ τη Βοσνία και ε, να διατηρήσει ένα περιβάλλον ασφάλεια ε, στην περιοχή. Η στρατηγική αναθεώρηση παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο στα κράτη-μέλη και είπαμε ότι πρέπει να περάσουμε από τη λογική του Dayton στη λογική των Βρυξελών. Θέλουμε να αξιολογήσουμε το ρόλο ε, των δυνάμεών μας ε, στην χώρα και στην, στην περιοχή γενικότερα. Δώσαμε έτσι μια νέα εικόνα για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι νέες δυναμικές στη Βοσνία Ζεγοβίνη στα πλαίσια της στρατηγικής αναθεώρησης, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν κάποιες προσαρμογές. Στην επιχείρηση συμφώνησαν ότι η στρατιωτική παρουσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει απαραίτητη, μια και η επιχείρηση Αλθέα παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για να βοηθήσει στο να εξασφαλίσει ένα ασφαλέ περιβάλλον. Συμφωνήσαμε ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στα βασικά μα καθήκοντα. Ε, Βεβαίω, ε, κάποιε άλλε επικουρικέ ε, επικουρικά καθήκοντα μπορούν να αναθεωρηθούν. Θα πρέπει να γίνουν κάποιες προσαρμογέ ε, για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να μπορούμε να βοηθήσουμε τις αρχές της Βοσνίας ε, να διατηρήσουν αυτό το ασφαλές περιβάλλον και να του δώσουμε τη δυνατότητα να επικεντρωθούν ε, στον δρόμο της ένταξης. Οι προσαρμογέ αυτέ θα εξηγηθούν πιο λεπτομέρω από τον συνάδελφο τον κύριο Σαλό, από τον ΝΑΤΟ. Αυτή αυτή η προσαρμογή περιλαμβάνει ε, την, ε, το να σταματήσει η δημιουργία εντολοτήτων και η κατάρτιση ε, που δεν χρειάζεται πλέον για κάποιες δυνάμεις, να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση έτσι ώστε η U4 να μπορεί να, να παίξει το βασικό της ρόλο μέχρι να πει την ενεργοποίηση των δυνάμεων που βρίσκονται εκτός της χώρας ε, εφόσον επιδεινωθεί σημαντικά η κατάσταση. υπάρχει και το καθήκον που έχει να κάνει με τα όπλα και τα και την διατήρησή τους. Γίνεται μια προσπάθεια συνεχής από την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε η Βοσνία Ζεγοβίνη να είναι η υποψήφια χώρα ε, για ένταξη το 2019. Είναι κρίσιμο αυτό το έτος για τις μεταρρυθμίσεις για να δει, επιδείξει η χώρα αυτή ότι σημειώνει πρόοδο ε, στον δρόμο τον ενταξιακό. Βεβαίως ε, το, πιο, το, το πρώτο εμπόδιο το πρώτο σημαντικό τεστ είναι οι εκλογές του Οκτωβρίου έτσι ώστε ε, να, θα πρέπει να προσέξουμε εκεί να μην επιδεινωθεί η κατάσταση πλευρά ασφάλεια, να μην, να μην υπάρξει εθνικό διχασμό. Μετά τι εκλογέ ε, και εφόσον έχουμε μια νέα υποψηφιότητα, θα πρέπει να επαναθεωρηθεί και ο ρόλο μα. Αλλά α φτάσουμε πρώτα εκεί και θα δούμε. Τα κράτη-μέλη έχουν ήδη συμφωνήσει για μια μελλοντική στρατηγική αναθεώρηση τη επιχείρηση Αλθέα που θα υποβληθεί στα κράτη-μέλη στις αρχές του 2019 για να αξιολογήσουμε σε ποιο βαθμό η Βοσνία Ζεγοβίνη έχει προχωρήσει στον ενταξιακό αυτόν δρόμο. Να σας θυμίσω ότι η επιχείρηση Αλθέα είναι η μόνη ευρωπαϊκή επιχείρηση ε, που διέπεται από συγκεκριμένου διακανονισμού. Έτσι, λοιπόν, η επιχείρηση Αλθέα δεν παίζει μόνο, μόνο πολύ σημαντικό ρόλο για να υπάρξει μια προοπτική ενταξιακή τη Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφαλίζοντα την ασφάλεια είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα τη σύγκληση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωσης. Θα ολοκληρώσω εδώ την παρουσίασή μου. Αν έχετε ερωτήσει, είμαι στη διάθεσή σας. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριο Τσίγκλερ. Έχω και εγώ κάποιες διαφάνειες. Θα σας μιλήσω για την κατάσταση της ασφάλειας από την οπτική γωνία της Κομισιόν και τι κάνουμε σε θέματα ε, χρηματοδοτικής στήριξης, αλλά όχι μόνο. Στην στρατηγική και τα Δυτικά Βαλκάνια που πρόσφατα υιοθετήσαμε, η Κομισιόν ε, ενισχύει τη στρατηγική συνεργασία ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικών Βαλκανίων. Είναι κάτι κέριο για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις υπάρχουσες απειλές που υπάρχουν για την Ένωση στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Φυσικά αποκλείεται να είναι αποτελεσματική ασφάλεια στα Δυτικά Βαλκάνια αν δεν εφαρμόσουμε το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία και αν δεν ενισχύσουμε την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταλήξει σε διάφορες εμβληματικές πρωτοβουλίες ε, για να αντιμετωπίσει τα διάφορα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν τα Δυτικά Βαλκάνια αποτελεσματικά και στο σύνολό τους ειδικότερα για τη Βοσνία Ζεγοβίνη, η προετοιμασία της γνωμοδότησης της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, αίτηση προσχώρησης της ε, Βοσνίας Ερζεγοβίνης που ζήτησε το Συμβούλιο από την Κομισιόν προσφέρει περαιτέρω ευκαιρίες για ανανεωμένη δεσμεύση σε διάφορους τομείς ασφαλείας και ειδικότερα στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και τη ριζοσπαστικοποίηση. Πολλά γίνονται ήδη όλες οι μεταρρυθμίσεις που υποστηρίζουμε μέσω της ενίσχυσης του κράτους δικαίου, ε, της αύξησης της αντοχής ε, στις απειλές ασφαλείας ε, θα μας βοηθήσουν. Να σας περιγράψω εν συντομία την τρέχουσα κατάσταση γιατί στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την πρόληψη του ακραίου εξτρεμισμού στη Βοσνία Ερσεγοβίνη. 118 άνθρωποι με την υπηκότητα τη Βοσνία Ερζεγοβίνης πιστεύετε, σύμφωνα με στοιχεία, ότι έχουν ταξιδέψει στη Συρία και το Ιράκ, άνδρε και γυναίκε. και από τη διασπορά ε, μεταξύ του 2013 και 2015. Οι αρχέ τη Βοσνία Ερζεγοβίνης έχουν καταβάλει προσπάθειε οι οποίε συνέβαλαν και πρέπει να το υπογραμμίσουμε, συνέβαλαν στο να, αναχαιτιστεί, να αναχαιτιστούν οι αναχωρήσει από το 2016 και μετά, σύμφωνα με πληροφορίε που έχουμε λάβει. Έχουν σταματήσει δηλαδή τέτοιε κινήσει από το 2016. Ε, Πυρήνε ριζοσπαστικοποίηση έχουν εντοπιστεί σε διάφορα σημεία ε, στη χώρα, ειδικότερα στι κοινότητε Βαχαμπή. Πολλοί άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν επιστρέψει ήδη και ο αριθμός ε, των επαναπατριζόμενων είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι και γυναίκε και παιδιά και δεν υπάρχουν υποψίες για εγκλήματα, αλλά κάποιοι έχουν ερευνηθεί και δικαστεί για τρομοκρατικά εγκλήματα. Έχουν λοιπόν ε, δοθεί όμως αποδοθεί συχνά ε, δικαστικές αποφάσεις ε, πολύ ήπιες λόγω έλλειψης στοιχείων. Υπάρχει ένας νόμος στη Βοσνία Ζεγοβίνη που λέει ότι αν κάποιος πρέπει να εκτίσει ποινή φυλάξη λιγότερη των νοσέτους, αυτή μπορεί να μετατραπεί σε πρόστιμο, σε χρηματική ποινή και αυτό τώρα έχει αλλάξει. Αυτή η μετατροπή σε ε, χρηματική ποινή έχει αλλάξει. Σε κάποια μέρη της χώρας και άλλα μέρη της χώρας συνεχίζουν να το κάνουν. Στη σερβική πλευρά και τώρα αρχίζει να εφαρμοστεί και στο υπόλοιπο της χώρας. Έχουν επιστρέψει διάφοροι, όπως είπαμε, πολίτες, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά. Ε, βασικές δυσκολίες ε, είναι η επανένταξη των αλλαδαπών μαχητών και η πρόληψη διαφόρων μορφών βίου εξτρεμισμού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε ένα ευαίσθητο ε, πλαίσιο όσον αφορά την εθνικιστική ρητορική που συχνά παρατηρούμε στη Βοσνία, ειδικότερα τους μήνες πριν από τις εκλογές. Εξού και ανάγκη ενίσχυσης του συντονισμού σε διάφορα θεσμικά επίπεδα διακυβέρνηση ώστε να υλοποιηθεί η σημερινή στρατηγική ε, καταπολέμηση τη τρομοκρατίας και του βιοεξτρεμισμού και μεταξύ των αρμόδιων ε, θεσμών στη Βοσνία Ζεγοβίνη και μεταξύ των εταίρων της στην περιοχή. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στον τομέα. Μέσω της συνεργασίας ε, πιστεύουμε ότι θα δοθούν αποτελέσματα. Αυτό που δεικνύεται από την ε, επίσκεψη που είχαμε ανώτων αξιωματούχων ε, στο Σεράγεβο πριν από ένα χρόνο για τα θέματα της αντιμετώπισης της δημοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού. Υπήρξαν ε, διάφοροι ανώτατοι αξιωματούχοι και ο δικός μας Γενικός Διευθυντής Ποπόφσκι και εκπρόσωποι από την DG Home. Ανώτατοι αξιωματούχοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση έκαναν διάφορες συστάσεις, παρότριναν τις αρχές ειδικότερα να ενισχύσουν το στρατηγικό πλαίσιο, την πρόληψη του βιοεξτρεμισμού, την ποινική δίωξη και την κράτηση αλλοδαπών μαχητών, την επιβολή του νόμου, συνεργασία με την Ευρωπόλ και την Eurojust, την καταπολέμηση του ξεπλήματο βρώμικου χρήματο και του παρανόμου εμπορίου πυροβολών όπλων. Ένα χρόνο μετά από την επίσκεψή του, η Κομισιόν ξεκίνησε μια συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και τον συντονιστή, τον αντιτρομοκρατικό συντονιστή, για θέματα αντιμετώπισης της τρομοκρατίας ε, και του βίαιου εξτρεμισμού. Αυτή την εβδομάδα πέντε εμπειρογνώμονες ε, δικοί μας βρίσκονται στη Βοσνία Ζεγοβίνη για να αναθεωρήσουν τι κάνουν οι αρχές για την υλοποίηση των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εμπειρογνώμονες ειδικότερα αξιολογούν, όπως βλέπετε, το στρατηγικό πλαίσιο και τις επιχειρησιακές δυνατότητες του δικαστικού των υπηρεσιών πληροφοριών και των αστυνομικών υπηρεσιών στο, στο αυτούς της ε, τρομοκρατίας και του βιοεξτρεμισμού. εξετάζουν διάφορες περιπτώσεις που αφορούν το κράτο δικαίου, από τι έρευνε μέχρι την επιβολή του νόμου, βελτιώνουν τη συνεργασία με διεθνεί εταίρου και άλλε χώρε στα Δυτικά Βαλκάνια. Αυτή η αποστολή επίση συμβάλλει σε έναν έλεγχο τη κατάσταση ε, των αντιδράσεων ε, των αρχών ε, βάσει απαντήσεων σε ένα ερωτηματολόγιο με πολλές ερωτήσεις που στείλαμε εμείς στη Βοσνία Ζεγοβίνη ε, είχαμε 20.000 σελίδες απαντήσεων που αυτή τη στιγμή μελετάμε ε, αφορούν τον τομέα της καταπολέμησης τρομοκρατίας και αυτοί, αυτές οι απαντήσεις μας δίνουν μια εικόνα της πραγματικής κατάστασης. Οι, οι διάφορες μέθοδοι καταπολέμησης τρομοκρατίας και του βιοεξτρεμισμού τι γίνεται με την ασφάλεια και το κράτο δικαίου. Όλα αυτά θα είναι στο επίκεντρο της δουλειά της Κομισιόν. Ε, ταυτόχρονα αυξάνουμε τη χρηματοδοτική μα στήριξη. Εντάσσουμε την αντιμετώπιση του βιοεξτρεμισμού σε όλα τα προγράμματα και στα τρέχοντα προγράμματα. Υπάρχουν 10 προγράμματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή ε, τα οποία συμβάλλουν για την ε, αύξηση τη αντοχή τη ε, απειλή ασφαλεία. Υπάρχει ένα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω για την ειρήνη και για την πρόληψη των κινδύνων ε, και το παράνομο εμπορίου. Το Συμβούλιο τη Ευρώπη υλοποιεί με δικά μα χρήματα ένα πρόγραμμα ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για του κρατούμενου και του κατα... κατάδικου. Επίση, χρηματοδοτούμε ένα έργο για τη ριζοσπαστικοποίηση σε φυλακέ και τρέχει επίση ένα πρόγραμμα στη Βοσνία ριζεγοβινη για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Όλα αυτά σε συνεργασία με την Ισλαμική Κοινότητα της ε, Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Επίσης, 13 είναι τα σχετικά περιφερειακά προγράμματα για όλη την περιοχή. Ένα από αυτά είναι η ανάπτυξη αξιωματούχων συνδεσμών της Ευρωπόλ στην Βοσνία Ερζεγοβίνη. Για να κλείσω, να σας πω ότι η Κομισιόν θα συνεχίσει να, στενά, να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον τομέα και να παρέχει περαιτέρω ε, οδηγίες ε, και καθοδήγηση στις αρχές ε, ώστε να αντιμετωπίσουν τις κοινέ προκλήσεις που θέτουν η τρομοκρατία και ο βίος εξτρεμισμός εκεί και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που βλέπετε στη διαφάνεια, αυτό είναι ένα από τα πράγματα που αναφέρθηκαν, το πλαίσιο Dayton, το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα δυσκολία ε, συνεργασία, ε, θέματα διακυβέρνηση και άλλα τέτοια ζητήματα. Αυτό είναι τα προβλήματα σε μια αποκεντρωμένη χώρα. Πάντα είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλά ειδικά στη Βοσνία Ζεγοβίνη είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολο να υπάρξουν κάποιε συμφωνίε με του αξιωματούχου συνδέσμου ε, σε ποιο σημείο πρέπει να γίνουν βελτιώσει. Αυτό θα βελτιωθεί στη διαδικασία αυτή τη προσχώρηση, ελπίζουμε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο σαν στον αντιστοματάρχη κύριο Νίκολα Σαλό, ο οποίος είναι στρατιωτικός επίκουρος του Δησασόρ. Ε. Γνωρίζετε πως παίζει ένα ιδιαίτερο ρόλο σε ό,τι αφορά και την ευρύτερη περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, οπότε η δική του παρέμβαση ε, θα είναι εξαιρετικά σημαντική. Τον ακούμε λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σωτήμα μέλη του Επιτροπής, στη και μετά την απόφαση του ΝΑΤΟ ε, στην ε, διάσκεψη κορυφής ε, της Κωνσταντινούπολης του 2004 να ολοκληρώσει την αποστολή S4 έως το 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε τη δική της αποστολή, την U4 αλθεα δηλαδή, με 2.000 προσωπικών. Ε, προσπαθώντας έτσι να εφαρμόσει τους όρους ε, της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του Dayton. Εδώ βασίζεται στην εκτελεστική εντολή που έχει λάβει, αλλά και στο ε, κεφάλαιο 7 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Στην τέταρτη έκθεση που δημοσίευσε τον Ιούλιο του 2017 το Ίδρυμα για τις Μελέτες Ασφαλείας Τη ε, Ευρώπη, ε, έθεσε το ερώτημα του τι θα συνέβαινε αν κατακαιρματιζόταν η ε, Βοσνία Ε, περιγράφεται δηλαδή εδώ ένα καταστροφικό σενάριο όπου ένα τμήμα της χώρας αποσκίζεται χωρίς με κάποιο ζήτημα των Ηνωμένων Εθνών να επιληθεί αυτό το ζήτημα. Ε, σε αυτό το σενάριο ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που θα οδηγούσαν σε αυτή την απόσχεση ε, εξωτερικοί παραγόντες οι οποίοι ε, ασκούν επιρροές στον πληθυσμό ε, δημιουργώντας, βασιζόμενοι μάλλον στην δύσκολη κοινωνικονομική κατάσταση και επιτείνοντας τις εθνικές εντάσεις. Εδώ έχει ληφθεί υπόψη και η ρίζοσπαστικοποίηση ε, του, ε, ε, της Ισλαμικής κοινότητας της Βοσνίας Ζεγοβίνης αλλά δεν υπήρχε και κατάλληλη πρόσβαση σε πληροφορίες σε ό,τι αφορά την ριζοσπαστικοποίηση και κατά συνέπεια την πρόληψή της. Επίσης δεν έχει υπάρξει σε αυτό το σενάριο η κατάλληλη ενημέρωση σε ό,τι αφορά τα πλεονεκτήματα από την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι με βάση τα στοιχεία τα πραγματικά που έχουμε σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση της Βοσνίας Ερζεγοβίνη προς την Ευρώπη. Γιατί αυτή τη στιγμή η κατάσταση παραμένει ήπια και δεν υπάρχει κάποια απειλή σε ό,τι αφορά το περιβάλλον ασφαλείας. Όμως είναι φυσικό και αναμενόμενο οι αρμόδιοι για την ασφάλεια να υπολογίζουν με τα χειρότερα ε, σενάρια. Υπάρχουν δηλαδή λόγοι ανησυχία και οι δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί θα πρέπει να είναι προετοιμασμένε. Ε, τον Οκτώβριο για παράδειγμα ε, του 2017 υπήρξαν ε, και εντάσεις και μεταξύ διαφορετικών εθνικότητων και ο πληθυσμός είναι εκνευρισμένος με το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη πρόοδος. Ναι, τα γενικότερα μακροοικονομικά στοιχεία βελτιώνονται, αλλά δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στην καθημερινή τους διαβίωση. Και η παρουσία και ενόπλων δυνάμεων εκτός των κανονικών ε, δομών δημιουργεί ε, περαιτέρω ανησυχία στο κοινό, ειδικότερα στη Ρεπούμπλικα Σύρψκα, καθώς δεν είναι ε, και γνωστό ποιος, ποιες ακριβώς είναι οι δομές αυτών, αυτής της στρατιωτικής δύναμης. Επίσης, υπάρχει αυξημένο τρομοκρατικό ε, κίνδυνο στην ε, Βοσνία Ερζεγοβίνη, ο οποίο επιτείνεται από την επιστροφή των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών. Ίσως θα θυμόσαστε ότι το Φεβρουάριο του 2014, όπως βλέπουμε στις ε, εικόνες εδώ, ξεκίνησαν κάποιες αναταραχές και διαδηλώσεις στη Βοσνία Ζεγοβίνη που κατέδειξαν ε, ε, τα προβλήματα σε ό,τι αφορά το τι θα πρέπει να γνωρίζει η νευτική δυνατή της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί. Και γι' αυτό θεωρούμε πως ε, η πρόσφατη απόφαση που έλαβαν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της PSC, στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Φραντέν, για την επανεδρέωση της EU4 ε, μέσω αυτού του υπονομαζομενου eu EU4 Task ε, ήταν η σωστή απόφαση. Ε, κατά την τελευταία μας εξάμεινη αξιολόγηση της EU4 Althea αναφερθήκαμε στο γεγονός ότι έχουμε μια καλύτερη γνώση της κατάστασης σε ό,τι αφορά και το εμψυχολικό αλλά και τον εξοπλισμό μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε κυρίως 600 άτομα προσωπικού που βρίσκονται στο Σαράγεβο και μπορούν να ενισχυθούν και να μετακινηθούν αλλού εάν αυτό χρειαστεί. Επίσης έχουμε ένα δίκτυο από 17 ομάδες ε, παρατηρητών και ομάδες ε, σύνδεσης ε, που συμβάλλουν στην αύξηση της προβολής στο κοινό της EU4. Από το 2010 η επιχείρηση Αλθέα έχει εστιάσει στη δημιουργία ικανοτήτων, το capacity building, αλλά και την εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων της Βοσνίας Ερσεγοβίνης. Αλλά μετά από τις συστάσεις που έγιναν τόσο από ε, τις ε, πολιτικές και στρατιωτικές δομές, αλλά και από την πίεση, ε, έχουμε ξεκινήσει τη σταδιακή κατάργηση ή τερματισμό αυτών των δραστηριοτήτων εκπαιδευτικών από τον τέλος του πολέμου του 1995 έχουμε ακόμα ε, να παραμένουν σε αυτή τη χώρα μεγάλα πλεονάσματα σε πυρομαχικά και πυροβόλα όπλα. Ε, και αυτή την περίοδο υποστηρίζουμε τις ενόπλες δυνάμεις της χώρας να, να, να καταστρέψουν αυτά τα πυρομαχικά ε, που φτάνουν σε 7.000 τόνους τα πυρομαχικά και 50.000 τόνους τα πυροβολά όπλα μέσω ενός συστήματος ανακύκλωσης. Επίσης η U4 διατηρεί μέσω ακριβώς συμφωνίας των Dayton το δικαίωμα να παρακολουθεί, να επαγρυπνεί και να ελέγχει οποιασδήποτε, ε, ε, τέτοιες δράσεις και σε ό,τι αφορά την, τον εξοπλισμό με πυροβολαόπλα των στρατιωτικών δυνάμεων. Επίσης, ε, η άρση ναρκοπαιδείων ε, ανήκει στις ε, αρμοδιότητες της EU4, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το επίπεδο της παροχής συμβουλών και της σύνδεσης. Παρότι πάνω από 3.000 τετραγωνικά μέτρα από το 1996 έχουν καθαριστεί από ναρκοπαίδια, χίλια τετραγωνικά μέτρα ακόμα παραμένουν ε, ε, ε, στην χώρα, γύρω στο 2,2% ακόμα της, της συνολικής επικράτειας παρουσιάζει κίνδυνο και συνολικά παραμένουν 79.000 νάρκες στη χώρα. Και βέβαια υπάρχει και ζήτημα διαφθοράς σε ό,τι αφορά αυτήν την όλη η επιχείρηση, καθώς μόνο για την απομάκρυνση μίας νάρκης χρειάζονται 6.000 ευρώ η οριστική απομάκρυνση των ε, ναρκοπαιδίων θα έχει ολοκληρωθεί ε, σε 9 με 10 χρόνια και μέσω του ICSP και της χρηματοδότησής του υπάρχει περαιτέρω υποστήριξη μέσω και ε, ερευνητικού προγράμματος το οποίο θα ξεκινήσει αυτό το μήνα και θα τρέξει για δύο χρόνια. Θεωρούμε πως ε, αυτή η έρευνα, αυτό το project θα μειώσει τις ε, προκλήσεις και μέσω της νέας προσέγγισης της επόμενες άρσεις ναρκοπαιδίων η Βοσνία Ζεγοβίνη θα μπορέσει να μειώσει το μέγεθος της πρόκλησης και κατά συνέπεια στο 2025 να έχει απαλλαγή πλήρως από τα ναρκοπαίδια. Και εδώ υπενθυμίζω τον αφορισμό του Winston ε, Churchill ότι δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα από όσα μπορούμε να κάνουμε. Παρ' όλα αυτό θα πρέπει να θυμόσαστε όλοι ποιος είμαι και γιατί σας μιλάω. Όσους ε, λοιπόν εγώ στρατιωτικός ε, επίκουρος του κ. Σερς Έντουαρτ που είναι ο DSSR και ο οποίος ε, παραμένει ένας από τους ε, στρατιωτικούς ηθήνοντες, να σας πω ότι είναι και ο επιχειρησιακό υπεύθυνο σε ό,τι αφορά τη τη φορά Ελπίζω να σας παρέχα χρήσιμες πληροφορίες σε ό,τι αφορά την περίπλοκη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα στη Βοσνία και Ζεγοβίνη. Λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται ως προπόθεση για να επουλώσει τις πληγές της αυτή η χώρα και προκειμένου να επανοικοδομήσει τις ε, δημοκρατικούς ε, θεσμούς, νομίζω πως θα πρέπει να παραλάβουμε τα όσα είπε ο Βαλέντι Ίνσκο μετά από την 15η επέτειο από την υπογραφή της Συμφωνίας ε, του Dayton στις 18 Μαΐου του 2017. Είπε λοιπόν πως η U4 είναι μια σχετικά αυτή, δηλαδή χωρίς ιδιαίτερο κόστος, αλλά σημαντική αποστολή U4 για τη σταθεροποίηση σε αυτή την περιοχή των Βαλκανίων. Σας ευχαριστώ. Να θυμίσω στους, στα μέλη του πάνελ και στους ε, ευρωβουλευτές ότι είχαμε το προνόμιο να μιλήσουμε και με τον Σερ Έρβαρντ στο παρελθόν ε, και όπως ε, έχουμε αποφασίσει, όχι σε υψηλότερο επίπεδο βέβαια, ε, ήταν πρόταση των, των κινήτων συντονιστών που έγινε αποδεκτή από την ΑΦΕΤ στο διευρυμένο Προέδριο ότι στο δεύτερο εξάμεινο του 2018 θα γίνει ε, αυτή η συνάντηση και μετά θα έχουμε και την αποστολή εκεί Λοιπόν, τώρα μπορούμε να περάσουμε στις ερωταπαντήσεις. Ο κύριος Πιτσολά έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις. Είναι πάντα καλό να μαθαίνει κανείς έτσι τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Βεβαίω και είναι καλό και αναγκαίο τα Δυτικά Βαλκάνια και η Βοσνία Ριζεγοβίνη ε, ιδιαίτερα ε, να επανέλθουν στα σχέδια τα ευρωπαϊκά διότι εξελίξεις από το 2014 στο 2018 δεν βοήθησαν και τόσο ε, ε, τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων δεν υπήρχε κάποιο όραμα για το μέλλον των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικών Βαλκανίων. Τώρα υπάρχει ένα πλαίσιο. Βεβαίως ε, μπορούμε να αναλύσουμε τι μπορεί να περιμένει κανείς ε, από αυτήν την στρατηγική ε, της μελλοντική διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως ε, υπάρχουν μια σειρά αποζητήματα, ε, όπως τα ζητήματα ασφάλειας βέβαια, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, και ένα από τους λόγους από τους οποίους ο κ. Γιούνκερ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησαν τη στρατηγική αυτή ήταν ε, το θέμα της ασφάλειας. Διότι τα Δυτικά Βαλκάνια εμφανίστηκαν στην πολιτική συζήτηση ε, όταν κυνηγούσαμε τους πάνωμους μετανάστες ε, και όχι πριν. Πλέον οι Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν ότι είναι το υπαριθμόν ένα ζήτημα η ασφάλεια και όχι τα οικονομικά και τα κοινωνικά. Βεβαίως ε, αυτό μας παραπέμπει στη σημερινή συζήτηση. Εμείς αναμένουμε με υπομονησία την επισκεψή μας ε, στη Βοσνία Ζεγοβίνη σε 15 μέρες. Ε, ήμουν εκεί πριν από 2,5 χρόνια, στα τέλη του 2015 και ε, πραγματικά θα πρέπει να δούμε ποια είναι η κατάσταση τώρα μετά από 2,5 χρόνια. Το εράτημά μου έχει να κάνει ε, με την ιδιότητά μου ως επικεφαλής της ε, αποστολή στο, στην Βοσνία Ζαβαβίνη και στο Κοσμοπέδιο δεν τέθηκε ποτέ το σύντημα της ε, αποστρατικοποίησης και νομίζω πως ήταν μια σωστή απόφαση διότι οι στρατιωτικές δυνάμεις πάντα δείχνουν είναι ένα στοιχείο μάλλον της ύπαρξης ενός κράτους και πρέπει να μπορεί να γίνει αυτή η επίδειξη ενός κράτους. Τώρα ποιες είναι αυτές δυνάμεις είναι άλλο ζήτημα. Οι στρατιωτικές δυνάμεις της Βοσνίας Ερζεγοβίνης είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος ε, και της δημιουργίας ε, μέτρων ε, οικοδόμησης εμπιστοσύνης διότι είναι κάτι που λειτουργεί είναι σημαντικό αυτό έχει ξεπεράσει και κάποιες προσδοκίες μπορεί η αστυνομία να μην λειτουργεί τόσο καλά αλλά οι στρατιωτικές δυνάμεις παίζουν το ρόλο τους από τότε που έχουν θεσπιστεί. Είναι σημαντικό λοιπόν να υποστηριχθούν οι στρατιωτικές δυνάμεις του Κωνσταντίνα Ε, τα ερωτήματά μου τώρα είναι ότι εξακολουθούμε να έχουμε 22.000 τόνους ε, ε, πυρομαχικών σε 17 διαφορετικά σημεία είναι σημαντικό το θέμα του στρατιωτικού υλικού που είναι αποθηκευμένου. Ε, η παρούσα κατάσταση στη χώρα επηρεάζει, την κατάσταση, επηρεάζει τα πράγματα ε, διότι όπως ξέρουμε είναι τοπικής διοκτησία αυτά τα πράγματα. Τι γίνεται λοιπόν με το θέμα αυτό της αποθήκευσης των πυρομαχικών. Θα ήθελα να ξέρω επίση τι γίνεται σε ό,τι αφορά το σχέδιο δράση για την ένταξη τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Θέλουν οι Βόσνοι να ενταχθούν. Ε, υπάρχουν όμως κάποιες φυλάξεις από την πλευρά του ΝΑΤΟ. Ε, υπάρχει μεταξύ άλλων το θέμα της στρατιωτικής ε, ιδιοκτησίας. Υπάρχουν μια σειρά από πολιτικά εμπόδια που τίθενται κυρίω από τη σερβική πλευρά. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω τι να πείτε και από αυτό Και το τελευταίο μου ερώτημα, την πρόσφατη, η πρόσφατη αγορά ε, αυτόματων όπλων ε, από την δημοκρατία, από τις αστυνομικές δυνάμεις της Ρεπούμπλικα Σέρβσκα, των Σέρβων της Σερβικής δηλαδή, Πώ το βλέπετε αυτό. Είναι κάτι που μπορεί να βελτιώσει την ασφάλεια στην περιοχή ή αντιθέτως ε, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Έχουμε και τις εκλογές που έρχονται. Δεν θα είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ε, ρητορικά θα ακουστούν έτσι αρκετά ακραία πράγματα. Είναι γνωστό το ιστορικό. Λοιπόν, άλλο πράγμα είναι να έχουμε στρατιωτικές δυνάμεις οπλισμένες και άλλο να ε, οπλίζουμε την αστυνομία μήπως ε, ε, αυτό θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από ότι οτιδήποτε άλλο. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιώσεφραντος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του πάνελ για τις παρουσιάσεις τους. Πιστεύω ότι η στρατηγική διεύρυνση που υιοθετήθηκε πριν από ένα μήνα και ειδικότερα το σχέδιο δράση, μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στις ε, προσπάθειες σταθεροποίηση στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Ωστόσο, η χώρα έχει να αντιμετωπίσει διάφορα πολιτικά προβλήματα. Αναφερόμαι και στον εκλογικό νόμο και στη διεξαγωγή πραγματικά δημοκρατικών εκλογών οι οποίες θα συμβάλλουν στη σταθερότητα της χώρας και στην πορεία της ε, για να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στρατηγική και το σχέδιο δράσης, τα οποία έχουν, προσφέρουν πολλές δυνατότητες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, πέραν της Βοσνίας Ρεζεγοβίνης. Ήθελα να εστιαστώ στα ζητήματα ασφαλείας. Ε, αυτό είναι το βασικότερο θέμα της σημερινής συζήτησης. Ο κ. Πίτσουλα ανέφερε ότι αγοράστηκαν πάνω από 22.000 2.000 ε, ε, πυρομαχικά, τεμάχια πυρομαχικών από τις δυνάμεις της ε, Δημοκρατίας της Σερβίας, της Ρεπούμπλικας Σέρψκα. Είναι πάρα πολλά αυτά τα πυρομαχικά για τις δυνάμεις για τις οποίες προορίζονται. Οπότε αυτό μας δίνει λόγους ανησυχίας. Υπάρχουν και άλλες ε, απειλές προς την ασφάλεια από την Ρεπούμπλικα Σέρψκα. Ε, διάφορες νυχτερινές κινήσεις ε, ενοπλών ομάδων, παραστρατιωτικών ομάδων και επίσης έχουμε και μια άλλη παραστρατιωτική ομάδα που προέρχεται από τη Ρωσία, η οποία πραγματοποιεί το γύρο των επωνομαζόμενων Ρωσικών Βαλκανίων η οποία μάλιστα συμμετείχε και στους ορτασμούς ε, της επαιτίου της ε, Ρεπούμπλικα Σέρψκα. Αυτά μαζί με άλλα πολλά ζητήματα που επιβαρύνουν τη Βοσνία Ερζεγοβίνη όπως η ριζοσπαστικοποίηση, οι αλλοδαποί μαχητές που επιστρέφουν από παιδιά μάχη στην αλλοδαπή. Η Ρεπούμπλικα Σέρψκα λοιπόν στέλνει ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα δείχνει ότι έχει ισχυρές σχέσεις με τη Ρωσία, κάτι που είναι ανησυχητικό. Και η ερώτησή μου είναι, έχετε καθόλου επιπλέον πληροφορίες όσον αφορά τον εξοπλισμό των αστυνομικών δυνάμεων στη Ρεπούμπλικα Σερψικά και ποια είναι η άποψή σα για αυτή τη διαδικασία που τρέχει αυτή τη στιγμή. Φαίνεται να ε, ενισχύονται οι παραστρατητικές ομάδες ε, στη Ρεπούμπλικα Σερψικά Ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Έντ. Ε, ζητώ συγγνώμη που δεν το προφέρω σωστά το όνομά σας, κυρία Πέτρη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, κύριε Μακάλιστερ, αγαπητά μέλη του πάνελ, συμφωνώ φυσικά με όλα όσα λέτε ότι η Βοσνία θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να τη βοηθήσουμε στη διαδικασία, να διατηρήσουμε τη Βοσνία Ζεγοβίνη ως μία χώρα, ενιαία χώρα, διασφαλίζοντας όμως και τα δικαιώματα των τριών λαών που την αποτελούν, κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα. Ωστόσο, είπα και κάτι άλλο σημαντικό. Θέλω να εκφράσω την ανησυχία μου για την κατάσταση όπως έχει αυτή τη στιγμή, ειδικότερα διότι εγώ ε, προέρχομαι από την Κροατία και η Κροατία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τα μεγαλύτερα σύνορα με την Βοσνία Ζεγοβίνη. Κατά μήκο των σύνορων αυτών εμφανίζονται διαρκώς ε, οικισμοί Ουαχάμπη και διάφοροι αλλοδαποί μαθητές επιστρέφουν σε αυτούς τους οικισμούς. Είχαμε και πολλές ε, περιπτώσεις όπου μετριοπαθείς ημάμιδες έκαναν έκκληση για για ε, ε, φιλική στάση προς το ευρωπαϊκό Ισλάμ και δέχτηκαν επιθέσεις και αυτοί και οι οικογένειες τους επίσης ε, παρατηρούνται, παρατηρείται να έρχονται χρήματα από χώρες οι οποίες είναι φιλικές χώρες προς την Βοσνία Ερσεγοβίνη μένα αλλά παρατηρείται κατάχρηση των χρημάτων αυτών παρέχονται υποτροφίες ε, μόνο εφόσον ας πούμε τα κορίτσια φορούν χιτζάμπ και μόνο αν οι άνδρες ε, έχουν ε, γενεάδα και τηρούν όλες τις θρησκευτικές τελετές διαφορετικά δεν παίρνουν υποτροφίες ως φοιτητέ. Αυτά τα χρήματα βοήθησαν να οικοδομηθεί και μια νέα πόλη την οποία κατοικεί αραβικός πληθυσμός. Βοσνοί σαλαφιστές. Φαίνεται να κλέβουν αυτοί οι άνθρωποι την ταυτότητα των πολίτων της Βοσνίας και αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα στους μουσουλμάνους. Διότι στην περιοχή αυτή ανέκαθεν υπήρχε συνύπαρξη, συμβίωση, αλλά σήμερα προωθούνται άλλες αξίες. Και θέλω να ρωτήσω τους ε, προσκεκλημένους μας και ειδικότερα τους ε, προσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρακολουθείτε τις ροές ε, αυτές ε, των χρημάτων που προέρχονται από τη Σαουδική Αραβία και από χώρες όπως η Τουρκία για παράδειγμα και από άλλες Ισλαμικές χώρες άλλες μουσουλμανικές χώρες οι οποίες ε, στέλνουν αυτά τα χρήματα στη Βοσνία Ερζεγοβίνη με σκοπό τη ριζοσπαστικοποίηση του πληθυσμού κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες απειλές ασφαλείας. Ευχαριστώ. Thank you, madam. I would like to, ask my questions as well. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κάνω και εγώ τις δικές μου ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα προς τον κύριο Τσίγκλερ και στον κύριο Φραντά. Θέλω να αναφερθώ σε ζητήματα δυναμικής ουσιαστικά ε, κινήσεων παρατηρούνται εντός της κοινότητας Βαχάμπη. Αυτή η διάδοση της ε, ε, φιλική στάση προς αυτή την ε, κοινότητα. Έχει ξεκινήσει εδώ και πάνω από 10 χρόνια νομίζω. Ήδη λοιπόν μας ανησυχούσε από τότε. Πώς αξιολογείτε εσείς ε, τη σημερινή δυναμική της διαδικασίας. Φυσικά αντιλαμβανόμαστε ότι γνωρίζουμε τις πηγές στήριξης Κάτι που είναι ανησυχητικό. Υπάρχει ανησυχία για τους αλλοδαπούς μαχητές που επιστρέφουν. Αλλά επίσης είναι ανησυχητικό ότι πηγαίνουν και τόσο πολλοί αλλοδαποί μαχητές στη Συρία από τη Βοσνία Ριζεγοβίνη. Κάτι που σχετίζεται με το γεγονός ότι υπάρχουν ριζοσπαστικοποιημένες βαχαμπιστικές ε, κοινότητες ε, εδώ και πολύ καιρό. Τόσο η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση όσο και η Κομισιόν λαμβάνουν υπόψη και παρακολουθούν στενά αυτέ τις δραστηριότητες. και για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση ε, των ανθρώπων και το συγχαίρω γι' αυτό. Η ερώτησή μου και προς τον κύριο Σαλόν αναφέρατε μία απόφαση σταδιακής ε, κατάρριξης της δραστηριότητας εκπαίδευσης της U4 Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα σχέδια για τις μελλοντικές ε, δράσεις, ποια είναι η αρχιτεκτονική, τι απαιτείται περισσότερο και ποια είναι τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να ληφθούν ώστε να ενισχυθούν οι ενόπλες δυνάμεις της Βοσνίας Αρζεγοβίνης. Θα ήθελα να μου πείτε και τη δική σας αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά την υλοποίηση συμφωνίας των Dayton και υπάρχουν δυνατότητες να επιταχυνθεί. Η εντολή ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να, να επηρεαστεί το πολύ τεταμένο πολιτικό περιβάλλον στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Εγώ ανησυχώ για την προεκλογική περίοδο. Επίσης όλα αυτά που ακούμε για τις παραστρατιωτικές ομάδες στην Ρεπούμπλικα Σέρψκα μου θυμίζουν τα πρώιμα στάδια του πολέμου στην Ουκρανία και το πολύ μεγάλο, πολύ ψηλό ενδεχόμενο αποσταθεροποίησης λόγω τέτοιων δραστηριοτήτων υβριδικού πολέμου. Το επόμενο μας σημείο μάλιστα αφορά τις θετικές επικοινωνίες. Ε, είναι πολύ σχετικό φυσικά. Αλλά αυτές οι παραστρατιωτικές ομάδες είναι πολύ δραστηριές και δημιουργούν ανησυχία. Να δώσω το λόγο στα μέλη του πάνελ με την ίδια σειρά. Ο κ. Φρέντο πρώτος. Thank you very much for... Σας ευχαριστώ πολύ για αυτά τα ερώτηματα. Θα αναφερθούμε στα ζητήματα ασφάλειας και άμυνας. Και εδώ θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως η Βοσνέζα Ζαγοβίνη είναι βρίσκεται σε ένα καθεστώς ε, ιδιαίτερα δύσκολο και όταν εξετάζουμε το μέλλον και ταυτόχρονα είναι μια υποψήφια προς προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα. Οπότε, όπως αναφέρθηκε, είναι εξαιρετικά σημαντικό και κρίσιμη σημασία σε σημερινή κατάσταση να περιγράψουμε τα πράγματα κάπω απεσιόδοξα ακόμα και όταν προσπαθούμε να είμαστε αισιόδοξοι και να έχουμε κάποια ελπίδα σε ό,τι αφορά αυτή την προσχώρηση στο μέλλον και το γεγονό ότι αυτή θα δημιουργήσει την απαραίτητη βούληση στην πολιτική ηγεσία για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα. Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ασφαλεία τώρα και το τι ακριβώ χρειάζεται αυτή η χώρα, χρειάζεται περισσότερη συνομία, χρειάζεται περισσότερε ένοπλε δυνάμει. Ε, αυτό εξαρτάται από τις απειλές που αντιμετωπίζει αυτή η χώρα. Ποιες είναι οι απειλές της, είναι εξωτερικές απειλές. Δηλαδή επιρροές από τρίτους παράγοντες, είναι εσωτερικές οι απειλές που προκύπτουν από το σύνταγμα της χώρας και το ότι δεν μπορεί δηλαδή να ενοποιηθεί ως έθνος. Ίσως έχουν ε, θρησκευτικό χαρακτήρα αυτές οι απειλές. Οπότε αφού αξιολογήσει, αφού αναγνωρίσει κανεί τι απειλέ, τότε μπορεί να γνωρίζει και τι είδου δυνάμει αστυνομικέ ή ενόπλε χρειάζεται. Και εδώ το ερώτημα σε ό,τι αφορά τη UFOR είναι αποτελεί ο στρατός ένοπλες δυνάμεις την απάντηση για τις απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα. Η αστυνομία αποτελεί λύση, αποτελεί ένα τμήμα στις λύσεις η αστυνομία, αλλά Ε, εκείνο πάντως που αποτελεί το συνδετικό ιστό της χώρας δεν είναι οι ένοπλες δυνάμεις, ε, ούτε η αστυνομία, είναι τα θεσμικά όργανα, ένα κοινό όραμα και η ελπίδα. Και θα πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου όταν θέλουμε να ορίσουμε το ποιος τελικά θα πρέπει να έχει εδώ την, ε, την, τις σχετικές εξουσίες στη Βοσνία Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ένοπλες δυνάμεις, να πούμε ότι εδώ πρόκειται για την αρχαιότερη, αν θέλετε, την παλαιότερη ε, αποστολή στο πλαίσιο κοινή πολιτική άμυνα και ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο Δημοτάρχη ε, Σαλόν μπορεί ενδεχομένω ε, μπορεί να επεκταθεί λίγο περαιτέρω πως για μας το ζήτημα δεν ήταν απλώς μόνο η υποστήριξη που παρήχαμε, εκτός και αν όλο αυτό το κομμάτι του CBNT περάσει και θεσμοθετηθεί περισσότερο. Άρα λοιπόν, Χρειαζόμαστε και περισσότερες αστυνομικές ε, δυνάμεις, αλλά τι είδους αστυνομικές δυνάμεις, και το αναφέρατε ήδη. Το να εξοπλίζουμε, για παράδειγμα, την αστυνομία με υπερβολικά πολύ εξοπλισμό, δηλαδή υπερβολικά πολλά όπλα, πέραν των όσων χρειάζονται ως αστυνομικές δυνάμεις, είναι κάτι που προκαλεί ανησυχία σε εμάς. Και τα κράτη-μέλη πραγματικά ανησυχούσιες με αυτό και νομίζω πως ο δικός σας εκπρόσωπος ε, στην πίεση το αναφέρθηκε σε αυτό όταν συζητήσαμε την εξάμεινη έκθεση της Αλθέα την περασμένη εβδομάδα. Άρα αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι πρόκειται εδώ για κάτι το οποίο παρακολουθούμε. Αλλά το ερώτημα εδώ είναι ε, τι είδους εξοπλισμό ε, εφοδιάζεται, με τι είδου εξοπλισμό εφοδιάζεται αυτή η αστυνομία, αλλά τι σκοπεύει να κάνει με αυτά τα όπλα, με αυτόν τον εξοπλισμό αυτή η αστυνομία. Και εδώ ακριβώ αξιώνουμε τη διαφάνεια που θα πρέπει να έχουν αυτές, αυτή η χώρα και οι δυνάμει ε, στο πλαίσιο ακριβώ τη πονταξιακής διαδικασία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι ε, μελλοντικέ εκλογέ και το περιβάλλον στο πλαίσιο που, που ε, αυτών των εκλογών, αλλά και το περιβάλλον μετά από αυτές τις εκλογές, είναι κάτι που μας προκαλεί ανησυχία. Ελπίζουμε δηλαδή πως θα λάβουμε χώρα ε, εγκαίρως ε, και σε, μια καλή ατμόσφαιρα, αλλά από εκεί και μετά τι θα γίνει είναι το ζητούμενο. Γιατί οι υποψήφιες προς προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες χρειάζονται μια τέτοια αποστολή, με εκτελετικού τύπου εντολή. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τοπική ανάληψη των ευθυνών δηλαδή από την κάθε χώρα, σε ό,τι αφορά την άρση των ανακοπαιδίων, σε ό,τι αφορά την καταστροφή των πυρομαχικών και πυροβολών όπλων, θα πρέπει να πούμε πω πραγματικά ε, δεν υπάρχει ένα όριστο όσο προσπαθεί να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τι ενόπλες δυνάμει. Σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα ζητήματα ε, ε, της ε, αποθήκευσης και ούτω καθεξής, αυτά μπορεί να σα τα διευκρινίσει ο κ. Σαλώνο, στρατιωτικό επίκουρο. πάντως ε, σε ό,τι αφορά τις ε, εκλογές ε, σε δημοκρατικό πλαίσιο προφανώς θα εξετάζουμε αλλά από εκεί και μετά σε ό,τι αφορά τα ζητήματα για παράδειγμα των θρησκευτικών τάσεων και των απειλών ή μάλλον τις αυξανόμενες επιρροής από αραβικές χώρες εδώ μπορώ να πω θα πρέπει να αξιολογήσουμε τη συγκεκριμένη απειλή σε σχέση και με τις υπόλοιπες. Έτσι ώστε να δούμε τελικά ποια είναι η σημαντικότερη απειλή για αυτή τη χώρα. Ελπίζω να απάντησα στα όλα τα ερωτήματα και τώρα να πάρει το λόγο λέει πρόεδρος ο κύριος ε, Τσέκλερ. Ε, ευχαριστώ να συμπληρώσω και εγώ κάπως ε, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, για ε, βεβαίως τα ξέρει πολύ καλά. Ε, θα ξεκινήσω με εσάς κυρία Φορτίγκα, σε ό,τι αφορά τα, τις βοχαμπιστικές οργανώσει. οργανώσεις. Ε, αυτές οι ομάδες είναι ουσιαστικά τα κατάλοιπα του πολέμου το 1995. Ε, είναι εκεί, είναι ένα πρόβλημα, παραδοσιακά η μουσουλμανική ε, κοινότητα στη Βοσνία Ζωκοβίνη είναι εξαιρετικά μετριοπαθής. Τώρα, αυτές οι Ισλαμιστικές ομάδες, ε, ο επικεφαλής εμπροσεπτός της μουσουλμανικής κοινότητας, ε, ουσιαστικά έστειλε ένα τελεσίγραφο σε αυτές τις ακραίες ομάδες να υπαχθούν ουσιαστικά στη μουσουλμανική κοινότητα. Δεν το έκαναν όλοι, ήταν 38 ομάδες και μόνο 14 μπήκαν ε, έτσι υπό την αιγίδα της Ισλαμικής κοινότητας, της μουσουλμανικής κοινότητας. Είναι δηλαδή άλλες 24 που είναι εκτός. Δεν θέλουν ε, να ε, υπαχθούν σε αυτό το μετριοπαθές Ισλάμ. Και αυτό είναι μια πρόκληση. Σε ό,τι αφορά τώρα τους ξένους μαχητές που φεύγουν από τη Βοσνία Ζεγοβίνη, αν δείτε τα συνολικά στοιχεία και να τα συγκρίνουμε, έτσι για να έχουμε κατά να, ξέρουμε και τι γίνεται. Ε, από το Βέλγιο ή από την Ισπανία. Ε, είναι πολύ περισσότεροι ξενιμαχητέ από το Βέλγιο από, από τη Βοσνία. Ε, από το 2016 δεν έχει γίνει καμία αναχώρηση. Δηλαδή υπάρχει μια σχετική ευαισθητοποίηση. Οι αρχές της Βοσνίας ε, έχουν ενημερωθεί, έχουν καταλάβει ότι είναι ένα ζήτημα εξαιρετικά σημαντικό για μας είναι και προτεραιότητα της κοινή γνώμης αυτό, οπότε αντιλαμβάνονται το πόσο σημαντικό είναι αυτό και για την ενταξιακή διαδικασία. Γι' αυτό έχουμε κάνει τι αποστολέ. Την αποστολή των εξόδων αξιωματούχων πέρυσι, έχουμε την αξιολόγηση ομορτήμων αυτή την εβδομάδα, ε, πιστολή, ε, αποστολή της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου, ε, του Κότερ, ε, θα πάτε κι εσείς. Όλα αυτά μας δίνουν την ευκαιρία να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση ε, εκεί και βεβαίω πρέπει να δούμε και τις ροές, τις χρηματικές. Ε, στο μέτρο του δυνατού το κάνουμε αυτό. Θα έχετε τη δυνατότητα να το δείτε όταν θα πάτε τη χώρα. Σε ό,τι αφορά τι παραστατιωτικέ ομάδε τώρα. Είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί Εάν πιστέψουμε τα μέσα ενημέρωσης ε, που είπαν ότι πριν από μερικά χρόνια υπήρχε μια παραστρατιωτική ομάδα εντός της Ρεπούλικας Σέρψκα όπου επικεφαλής ήταν ε, στο παρελθόν στην Ανατολική, ήταν μετά στην Ανατολική Ουκρανία στον Ντόμπας ε, αυτό δείχνει ότι εντάξει, υπάρχει ένα επίπεδο επικινδυνότητας και είναι κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου ευχάριστο, είναι μια απειλή, μια πρόκληση θα πρέπει όλα αυτά να τα παρακολουθούμε και θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν αυτό και οι αρχές. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν τώρα με τον χάρτη και που ε, βεβαίω ε, το ΝΑΤΟ υπεύθυνο, νομίζω ότι ο αντισταγματάρχης είναι σε καλύτερη θέση για να απαντήσει. Έχετε το λόγο κύριε Σαλό, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε πέντε ερωτήματα νομίζω αφορούσαν την ασφάλεια και δύο τις στρατιωτικές δυνάμεις της Βοσνίας και ε, για τις τις ομάδε. ομάδες ε, θα πρέπει να πάμε στην ιστοσελίδα της aljazeera.com εκεί υπάρχει ένα άρθρο πριν από 12 ώρες αναρτήθηκε που λέει είναι η Βοσνία, η Νέα, η νέα Ουκρανία αυτός είναι ο τίτλος από ό,τι φαίνεται υπάρχει μία ε, κίνηση για να δημιουργηθεί ένα αποσχιστικό κίνημα ε, από τους ε, Σερβοβόσνιους. Ε, υπάρχουν ανησυχίες ότι αυτές οι ενδυνάμει παραστηριοτητικές ομάδες ε, ε, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν. Θα πρέπει βεβαίως να δούμε ποια είναι η απόσταση ανάμεσα σε κάποιε ομάδε βετεράνων του πολέμου και μια πραγματική παραστρατιωτική ομάδα. Γι' αυτό λοιπόν ζητούμε να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στην επιχείρηση Αλθέα, στις δυνάμεις της UFOR. Η αξιολόγηση μα αυτή τη στιγμή για τι ομάδε αυτέ είναι ότι είναι δύσκολο να τις κρίνουμε, θα πρέπει να έχουμε πιο πολλά στοιχεία, να γνωρίζουμε ποια είναι τα δίκτυα, να δούμε πώς σχετίζονται και με πολιτικούς ε, ηθήνοντες, πολιτικά πρόσωπα. Είναι ανοιχτό το θέμα αυτό, εν πάση περιπτώσει. Τώρα για την αποστολή των αυτόματων όπλων. Όπως ελέγχθη νωρίτερα, αυτά αγοράστηκαν νόμιμα. Είναι κάπως δυσανάλογο το μέγεθος βέβαια, Εμείς έχουμε ένα όπλο για 10 αστυνομικού στις δυνάμεις μας, στην Ευρώπη και στην Ρεπούλικα Σέρψκα υπάρχει ένα αυτόματο όπλο για κάθε αστυνομικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, την εντολή που έχουμε από τον Dayton, ε, εμείς παρακολουθούμε αυτές τις αστυνομικές δυνάμεις. Υπάρχουν 16 διαφορετικές ε, ε, υπηρεσίες επιβολής του νόμου στη Βοσνία Ζεγοβίνη που χρηματοδοτούνται ξεχωριστά η COM-UFOR έστειλε μια επιστολή σε όλες αυτές τις αρχές ε, για να μας στείλουν το κατάλογο με όλα τα όπλα τους. Αναμένουμε σύντομα τις απαντήσεις και βεβαίως αν χρειαστεί θα γίνουν και επιθεωρήσεις για να επαληθεύσουμε ότι ο κατάλογος που θα μας στείλουν είναι και σωστός. Τώρα για τη ριζοσπαστικοποίηση και την επιστροφή των ξένων μαχητών. Ε, δεν είναι τα πράγματα εκτός ελέγχου, δεν είναι δυσανάλογα σε σχέση με το τι γίνεται σε άλλες χώρες και ευρωπαϊκές χώρες. Βεβαίως παρακολουθούμε και τα οικονομικά δίκτυα αυτή τη στιγμή οι πιο ορατές επενδύσεις των χωρών ε, του κόλπου έχουν να κάνουν διακοπές, με θέρετρα παραθερισμού. Χρειαζόμαστε πιο πολλά στοιχεία σε επιπεδο να πούμε κάτι περισσότερο από αυτού για τα πυρομαχικά και ε, τα εκρηκτικά, AWE όπως τα ονομάζουμε, η τελευταία αξιολόγησή μας είναι ότι υπάρχουν 7.000 τόνοι πλεόνασμα χρειάζεται και 8.000 τόνους για τη χρήση τους δηλαδή μιλάμε για 15.000 τόνους συνολικά πυρομαχικών και εκρηκτικών στη Βοσνία Τσοκοβίνη η EU4 βοηθάει ε, τις ε, δυνάμεις της Βοσνίας για να διαχειριστούν αυτό το πλεόνασμα. Υπάρχει ένα master plan ε, μέσω του οποίου συντονίζουμε ε, τις δυνάμεις ε, της Αυτό γίνεται στα πλαίσια της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του Dayton και υποστηρίζουμε έτσι τις στρατιωτικές δυνάμεις της Βοσνίας. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να απαλλαχθούμε ε, από, αυτές, από αυτά τα πλεονάσματα έως το 2019 να είμαστε στο κατάλληλο επίπεδο έτσι ώστε να υπάρχει από ένα σημείο και μετά αυτάρκεια. Είμα, είναι, έχουμε δουλειά μπροστά μας, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το master plan για τα πυρομαχικά ε, και τα, ε, τα εκρηκτικά έως το 2019. Εμείς έχουμε δώσει την, ε, ε, τη συμβουλή στην Επιτροπή για την Ασφάλεια να συνεχιστεί έως το 2020 η εντολή για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις ε, στρατιωτικές δυνάμεις να μπορέσουν να ε, απαλλαγούν και από τα ελαφριά τους όπλα, περίπου 15.000, αναμένουμε απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό. Τώρα για τις εκλογές, ε, όπως είπα, εντάξει είναι κάτι που μας απασχολεί. Αναμένουμε και εδώ μια απόφαση για τα περαιτέρω ε, στοιχεία που ζητήσαμε στα πλαίσια της επιχείρησης Αλθέα ε, για την υπηρεσία πληροφοριών. Θα πρέπει πάντως να αυξηθεί η προσπάθεια ευαισθητοποίησης. Να σας πω ενημερωτικά ότι οι επιχειρησιακές ε, μάλλον πέντε εβδομάδες πριν για τις κοινικές εκλογές θα γίνει μια επιθεώρηση των δυνάμεών μας εκεί πρέπει οπωσδήποτε να αισθάνονται ασφαλείς οι πολίτες στη χώρα αυτή. Για τις στρατιωτικές δυνάμεις τώρα, πρώτα απ' όλα για το Membership Action Plan και ε, την κατάρτιση είναι πολιτική απόφαση το σχέδιο δράσης ε, για την υποψηφιότητα και το εμπόδιο είναι αυτή τη στιγμή οι προποθέσει του Τάλιν που λένε ότι πρέπει η Βοσνία ως κράτος να εγγραφεί και να καταγράψει όλα τα στοιχεία τα αμυντικά. Πάνω από 50% αυτών των περιουσιακών στοιχείων είναι καταγεγραμμένα όλα στην Ομοσπονδία ε, της Βοσνίας, αλλά τίποτα απολύτως από την Ρεπούμπλικα Σέρψκα, από τους Σερβοβόσνιους δηλαδή. Θα πρέπει από εκεί και πέρα να αποφασίσουμε εάν θα αφήσουμε μια οντότητα όπως η Ρεπούλικα Σέρψκα ε, να ασκήσει βέτο σε αυτό το σχέδιο το ή αν θα προσπαθήσουμε να εκμελευτούμε τη συγκυρία, ε, την πρόοδο που υπάρχει για να προχωρήσει το σχέδιο. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης ε, την οποία αναμένουμε. Γνωρίζουν το ζήτημα αυτό οι ευλεγόμενοι φορείς. και θα δούμε τι θα συμβεί, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Για την κατάρτιση ακολουθήσαμε τις συστάσεις ε, της ε, ομάδας πολιτικής ε, για να δούμε πώς κάποιες δράσεις κατάρτισης θα μειωθούν, κάποιες όμως μόνο. Η προσθέμενη αξία είναι η υποστήριξη του πολυεθνικού, των πολυεθνικών δυνάμεων, των στρατιωτικών, να τους βοηθήσουμε για να μπορεί να λειτουργεί στο σχέδιο διαλειτουργικότητας του ΝΑΤΟ, ε, να φτάσουν προς τα πρότυπα του ΝΑΤΟ που να τους επιτρέπει να στέλνουν επιχειρήσεις, ε, να στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις σε επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για ΝΑΤΟ, είτε μιλάμε για ε, Ηνωμένα Έθνη. Αυτή τη στιγμή περίπου 16 στρατιώτες συμμετέχουν σε επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και άλλες χώρες της Αφρικής. θα συνεχιστεί αυτή η υποστήριξη. Αυτή ήταν η συστασή μας, δεν μας κοστίζει και κάτι. Και οι στρατιωτικές δυνάμεις της Βοσνίας ελπίζουμε να αναλάβουν κάποιες ευθύνες, ε, να υπάρξει μια οικειοποίηση μέσω του, σχέδιου, του κέντρου κατάρτισης ε, που υπάρχει στο Σαράγεβο. Τώρα γιατί γιατί μπορούμε να μειώσουμε αυτές τις δράσεις. Μόλις 5-10% της κατάρτισης γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το υπόλοιπο γίνεται από τον ΝΑΤΟ ή μέσω διμερών συμφωνιών. Ε, οπότε εδώ έπαιξε ρόλο η συνεργασία ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζουμε το αρχηγείο του ΝΑΤΟ στο Σαράγεβο να βοηθήσει για τον συντονισμό αυτών των δράσεων κατάρτισης. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ. Πολύ κατανοητό. Ευχαριστούμε πολύ. Μιλήσαμε, πιστεύω, επαρκώς για αυτό το σημείο. Θα ακολουθήσει μάλιστα και ένα άλλο σημείο για τα Δυτικά Βαλκάνια να ευχαριστήσω τα αξιότιμα μέλη του πάνελ. Μία τελική παρατηρήση, ένα σχόλιο στη ΣΕΝΤΕ. Είμαστε πιο τεχνικοί εκφύσεως. Είναι τεχνικές ερωτήσεις. Μας θέλουμε να μάθουμε τις λεπτομέρειες κάθε προβλήματος. Ωστόσο, όπως αποφασίσαμε στους συντονιστές ομόφωνα, θα πάμε στη Βοσνία Ζεγοβίνη για δεύτερη φορά σε αυτή τη θητεία. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ελπίδα και ότι μας αφορά σε μεγάλο βαθμό η ασφάλεια αυτής της χώρας. Την υποστηρίζουμε τη χώρα αυτή στο ε, δρόμο προς την προσχώρηση. Οι συνομιλητές μας εδώ οι περισσότεροι, οι περισσότεροι ήταν, είναι μέλη της ε, κεντρικής, ε, ανατολικής και νοτιάς Ευρώπης. Όλοι αυτοί οι βουλευτές συνήθως υποστηρίζουν τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μας λείπει λοιπόν ελπίδα. Αντιθέτως, μας ενδιαφέρει η κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Το επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης εστιάζεται επίσης στα Δυτικά Βαλκάνια και πιο συγκεκριμένα σε ένα θέμα που ενδιαφέρει εμένα ιδιαίτερα τις στρατηγικές επικοινωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Δυτικά Βαλκάνια. Να καλωσορίσω τους τρεις διακεκριμένους ε, τα μέλη του πάνελ. Ο πρώτος ο κύριος Λουτς Γκόλνερ, ε, των στρατηγικών επικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ο κύριος Κλάους Γκίρινγκ. Ο κύριος Κλάους Γκίρινγκ από την DGNIR στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τμήματάρχης και τελευταίος ε, η κυρία Ρόζα Μπαλφόρ από το German Marshall Fund των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακούσαμε ε, εισαγωγικά πολύ σωστά ότι την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τους εκπροσώπους των ε, θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΝΑΤΟ για την κατάσταση ασφαλείας στη Βοσνία Ερζογοβίνη. Είχαμε και τον επικεφαλής της αποστολής που θα ξεκινήσει αμέσως μετά το Πάσχα στο Σεράγεβο και τον, ε, τον εκπρόσωπο της ε, Ιουλφορανθέα να δώσω πρώτα απ' όλα το λόγο στα μέλη του πάνελ. Ε, κύριε Γκόλνερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις δραστηριότητες μας σε αυτό το πολύ σημαντικό τομέα. Να τονίσω ότι οι σημερινές μας παρουσιάσεις έχουν γίνει σε συνεργασία με την Κομισιόν. Αυτό θέλω να τονίσω ότι δεν εργαζόμαστε ξεχωριστά, αλλά συνεργαζόμαστε στενά. Θα είμαι σύντομος. Θα σας παρουσιάσω κάποιες πτυχές της προσέγγισης που ακολουθούμε, το περιεχόμενο και μερικά λόγια για τη δομή. Οι στρατηγικές επικοινωνίες, ε, κατά την άποψή μας, πρέπει να δοθούν από ολιστική οπτική γωνία. Δεν είναι μόνο μέσα μαζική ενημέρωση και σχέση με τον τύπο, είναι μια ολιστική προσέγγιση. Πιστεύω θα τη βρείτε πολύ σωστή γιατί ευθυγραμμίζεται με την έκθεση του Οκτωβρίου του 2016. Αυτή η προσέγγιση μας. Πολλές πτυχές λοιπόν των επικοινωνιών από επαφή με πολλαπλασιαστές, με κοινό απευθείας, με δίκτυα, περισσότερο παρά μια μονόδρομη επικοινωνία από πάνω προς τα κάτω. Αντιμετωπίζουμε επίσης ζητήματα τα οποία δεν έχουμε ξανααντιμετωπίσει. Αφορούν την παραπληροφόρηση και την αντοχή αφετηρία είναι η στρατηγική που εθετήθηκε πρόσφατα. Δεν χρειάζεται να σας την παρουσιάσω, τη γνωρίζετε. Για μας είναι ένα σημαντικό στοιχείο που θα μας ε, δώσει νέα δύναμη ε, και ένα νέο αφήγημα όσον αφορά την προσέγγιση μας ε, των επικοινωνιών εδώ. Στις στρατηγικές μας επικοινωνίες θέλουμε να διασφαλίζουμε δημόσια στήριξη για τους στόχους που διατυπώνται στρατηγική βάσει δύο γραμμών. Πρώτον στην περιοχή με τον κόσμο εκεί στα Δυτικά Βαλκάνια αλλά και με το δικό μας κόσμο εδώ, εδώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύο ξεχωριστά ακροατήρια. Με την ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης έχουμε μια ειδική ομάδα για τα Δυτικά Βαλκάνια. Είναι μικρή, αλλά αναπτύσσεται. Αυτό μαρτυρά και το πόση σπουδαιότητα εμείς δίνουμε στο ζήτημα αυτό. Επικοινωνούμε για το γενικότερο ζήτημα της ευρωπαϊκής στήριξης που βασίζεται σε συγκεκριμένα πράγματα. Θέλουμε δηλαδή να δείξουμε στα Κροατήρια, στα Δυτικά Βαλκάνια, ότι οι δραστηριότητες μας, η υποστήριξή μας προς την περιοχή έχει μια πραγματικά θετική επίδραση στην καθημερινή του ζωή ότι δεν τους ε, επικοινωνούμε χαρτιά και διαδικασίες, αλλά πράγματα τα οποία έχουν σημασία για τους πολίτες, για τους λαούς. Έχουμε διάφορα παραδείγματα που θα παρουσιάσει και ο συνάδελφος μου Γκίρινγκ σε λίγο. Η συνολική προσέγγιση, επαναλαμβάνω, για μας εστιάζεται στο να δώσουμε ένα θετικό αλλά ρεαλιστικό μήνυμα για τις προοπτικές που παρέχει αυτή η διαδικασία που έχουμε ξεκινήσει. Δεν τους λέμε δηλαδή τι κάνουμε ακριβώς, αλλά γιατί είναι σημαντική αυτή η διαδικασία για τους πολίτες των Δυτικών Βαλκανίων και για τη δική μας πλευρά. Έχουμε αναλύσει διάφορα θέματα τα οποία παρουσιάζουμε. Ένα πολύ σημαντικό πολιτικό είναι η πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Κάτι που μας δένει ουσιαστικά μαζί, που είναι κοινό για όλους μας είναι ένα μείγμα ενός στοιχείου ήπιας ε, εξουσίας αλλά και ένα στοιχείο που μας δείχνει ότι ανήκουμε στον ίδιο κόσμο όλοι. Συνεργαζόμαστε στενά προφανώς με το δίκτυό μας, με τις δικές μας αντιπροσωπείς που παίζουν σημαντικό ρόλο στην περιοχή. Συνεργαζόμαστε όμως και με εταίρους ε, στην περιοχή θέλουμε να συνεργαζόμαστε με τις ίδιες κυβερνήσεις πρώτον, αλλά και με μη κυβερνητικές οργανώσεις της περιοχής. Και φυσικά και κάτι άλλο πολύ σημαντικό για μας είναι η στενή συνεργασία και τονίζεται αυτό το σημείο στην έκθεση του Οκτωβρίου του 2016. Θέλουμε να έχουμε πιο ε, προσέγγιση με μεγαλύτερη επαφή με τα κράτη-μέλη. Θέλουμε δηλαδή να συγκεντρώνουμε τους εκπροσώπους, τους αρμοδίους ε, επικοινωνίας ε, της περιοχής για θέματα προσχώρησης, ώστε να συναντιόμαστε όλοι μαζί να καθορίζουμε στρατηγικές προσεγγίσεις και συγκεκριμένες αυτές δράσεις. Το ζήτημα της παραπληροφόρησης φυσικά απασχολεί τους πάντες. Τι να κάνουμε στα Δυτικά Βαλκάνια. Αντλούμε από την εμπειρία που αποκτήσαμε από τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας, ειδικότερα με την σχετική task force που έχουμε, που, η οποία έχει μια πολύ σαφή εντολή, όπως γνωρίζετε, από το 2015. Συγκεκριμένα καθήκοντα που εστιάζονται στην ε, ε, κοινοποίηση των προσεγγίσεων και των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Αλλά αναφέρουμε επίσης και πώς υποστηρίζουμε το περιβάλλον των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην περιοχή και τέλος πώς ε, αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο της παραπληροφόρησης στην περιοχή. Τέλος, τους περιορισμένους πόρους που έχουμε τους διαθέτουμε κυρίως στην αξιολόγηση του εύρους και του βάθους της πρόκλησης. Θέλουμε δηλαδή να εντοπίσουμε τι αφηγήματα κυκλοφορούν και να δούμε πώς επηρεάζουν τις δικές μας δραστηριότητες ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θέλουμε να δούμε κατά πόσο οι δραστηριότητε μα, οι στόχοι μα εκπροσωπούνται επαρκώ και πιστεύουμε σε μια προενεργό προσέγγιση επικοινωνία παρά σε εκ των υστέρων ε, επικοινωνία. Αυτός πιστεύουμε είναι ότι ο καλύτερος τρόπος ε, να αντιμετωπίσουμε αυτά τα αφηγήματα της παραπληροφόρησης, να είμαστε συγκεκριμένοι, ε, ρεαλιστικοί, ορατοί, να έχουμε μεγάλη προβολή και να επισημαίνουμε την τεράστια συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή αυτή. Και όλα αυτά βάσει πραγματικών γεγονότων φυσικά. Το τελευταίο που θέλω να πω πριν δώσω το λόγο στον συνάδελφο μου για να συμπληρώσει, αφορά τις δομές. Όπως σας είπα, έχουμε μια ειδική task force στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για αυτό το τομέα, για αυτή την περιοχή. Πιστεύουμε στη στενή συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων από πλευράς κομισιών, κρατών μελών και κάτι άλλο που διερευνάμε είναι η συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών στα Δυτικά Βαλκάνια και με τις κυβερνήσεις βέβαια της περιοχής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Γκέριγκα από την DGNR της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ζητώ συγγνώμη που δίστασα. Ε, να πω το όνομά σα Είναι η δεύτερη μέρα που πρόεδρευα αυτή την υποεπιτροπή. Έχω... Μπορεί να αντιμετωπίσω μερικά προβλήματα και ευχαριστώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για αυτή την πρόσκληση και νομίζω πως ε, είναι η σωστή χρονική συγκυρία για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία μας με τα Δυτικά Βαλκάνια στο πλαίσιο και της νέας στρατηγικής για αυτές τις χώρες. Όπως ο Λούτσε ήδη ανέφερε, πρόκειται για μια κοινή δράση από πλευρά της Επιτροπής και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και το λέω της Επιτροπής ειδικότερα της Διανικής Διεύθυνσης ΝΙΑ ε, ε, ξεκινώντα από τι δομέ, όπω είπε και ο Λούτσε, έχουμε δημιουργήσει από κοινού με τη Γενική Διεύθυνση μία, μία μικρή ομάδα προκειμένου να έχουμε καλύτερη επικοινωνία με τι αντιπροσωπείε μα ε, όταν αφορά την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Ουσιαστικά δηλαδή <clears throat> έχουμε δύο ομάδε, μια βασική ε, ομάδα πυρήνα και από εκεί και μετά μια δεύτερη, αλλά όπως είπε και ο Λούτσε προσπαθούμε να μην ε, εργαζόμαστε μόνοι μας σε ένα θελάκα αποκλεισμένοι, αλλά ε, να έχουμε συνεχή επικοινωνία με τους διάφορους φορείς μας οι οποίοι υλοποιούν και τα διάφορα προγράμματα, για παράδειγμα οι οργανισμοί ανθρωπιστικής βοήθειας, ε, χρηματοδότηση επενδύσεων, τις ε, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ούτω καθεξής. Ένα από τα κυριότερα σημεία στα οποία εστιάζουμε, για παράδειγμα, είναι οι νεότερε γενιές δηλαδή οι νέοι αποτελούν προτεραιότητα. Και πλήσει στο πλαίσιο των διασκέψεων κορυφής στην Παρίσι και στο Τριέστε, ε, διοργανώσαμε και μια μεγάλη διάσκεψη νέων, όπου προσκαλέσαμε ακριβώ νέου από τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τι χώρε των Δυτικών Αλβανίων, προκειμένου να ανταλλάξουν βέλτιστε πρακτικέ και να ανταλλάξουν απόψει και το κάναμε αυτό τόσο σε επίπεδο της Γενικής Νέρα, αλλά και στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή ζητήσαμε το Κοινοβούλιο να γίνει μια παρουσίαση ε, των, της πρωτοβουλίας νέων ηγετών. Και από εκεί και μετά είχαμε και πέρσι μια διάσκεψη στα πλαίσια του ε, διαλόγου υψηλού επίπεδου με τα Δυτικά Βαλκάνια. Εκεί λοιπόν προσκαλέσαμε νέους πολιτικούς από όλες αυτές τις χώρες των Δυτικών Βαλκαλίων και τους φέραμε ε, σε επαφή με άλλους νέους από εδώ και με εκπροσώπους της ε, των νέων, προκειμένου της νεολαίας, για να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε περισσότερο την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οργανώσεις της νεολαίας προφανώς είναι πολύ σημαντικές ε, για μας προκειμένου να επιτείνουμε την συνεργασία μας ε, και υπάρχει και ένα γραφείο συνεργασίας με τις οργανώσεις της νεολαίας το οποίο συστάθηκε πρόσφατα. Επίσης, όπως ανέφερε ήδη ο Λούτς, διαφοροποιήσαμε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε. Από τότε δηλαδή που είχαμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου το 2015 ε, και την έκθεση της Τσέρ ε, το 2016, ε, αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να ε, όχι μόνο να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση, αλλά να ενισχύσουμε και τις ε, θετικέ ειδήσει, ε, δηλαδή να αυξήσουμε και την ήπια σχήμα στο soft power. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε πώ μπορούμε να αλλάξουμε τη στρατηγική μας και αντί να μιλάμε πλέον για project, να μιλάμε για ενημερωτικέ. ενημερωτικές. Δηλαδή να εξηγούμε το γιατί προβαίνουμε σε ανταλλαγή απόψεων με τις χώρες εταίρου, το ποια είναι τα πλέον εκτήματα και όταν κάνουμε την επικοινωνία δεν λέμε ποια είναι τα κονδύλια τα οποία θα πανούμε, αλλά ποια είναι τα αποτελέσματα, ποιο είναι ο συγκεκριμένος αντίκτυπος για τους ανθρώπους των προγραμμάτων μας. Αυτά είναι τα βασικά μηνύματα, αυτά είναι τα αφηγήματα, αν θέλετε, τα narratives ε, τα οποία προσπαθούμε να περάσουμε και προσπαθούμε να αυξήσουμε και τη σχετική ικανότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε έναν στρατηγικό διάλογο ε, με τον Επιτρόπο Χαν ε, και ο κ. Μαχάριστα συμμετείχε εκεί και είπαμε ότι θα πρέπει να αυξηθεί η ορατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε δηλαδή να επιτρέπουμε ε, τρίτες χώρες ε, και άλλες ε, περιοχές να θεωρούνται ως κύριοι χωρικοί στη Σερβία όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσε και αποτελεί εδώ και σειρά ετών και τον κύριο χορηγό και τον βασικότερο εμπορικό εταίρο της χώρας. Άρα λοιπόν πρόκειται για πραγματικά στοιχεία και γι' αυτό θα πρέπει να αλλάξουμε και τις αντίστοιχες εντυπώσεις που υπάρχουν σε αυτές τις χώρες. Οπότε θα πρέπει να δώσουμε και στα διάφορα project τα οποία ελοποιούμε μια σαφή ευρωπαϊκή ταυτότητα. Δηλαδή να λέμε στις διάφορες εκστρατείες Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενέργεια, Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιχειρηματικότητα. Έχουμε για παράδειγμα ε, μια εκστρατεία που έχουμε ξεκινήσει στην πρώην Δημοκρατία της Μακεδονίας ε, όπου λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση για την νεολαία. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουμε με απλά πράγματα όπως ο τίτλος τον οποίο δίνουμε στις δράσεις μας έτσι ώστε να αυξήσουμε την ορατότητα της ε, Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αλλάξουμε τελικά την αντίληψη του κοινού εκεί ως προς το ποιο είναι εκείνο ο οποίο προβαίνει σε τέτοια υποστήριξη. Τώρα, πώ το επιτυγχάνουμε αυτό. Προφανώς υπάρχει ένα συντονισμό ε, και κοινή διοργάνωση των δραστηριοτήτων εδώ στις Βρυξέλλες, αλλά από εκεί και μετά εκείνο που καλείται να κάνει τη δουλειά του outreach, να έρθει σε επαφή δηλαδή με τις διάφορες κοινότητες είναι οι ε, πρόσωποι μας εκεί. Γιατί βέβαια θα πρέπει να υπάρξει επαφή όχι μόνο με τις πρωτεύουσε αλλά και με τις κατατόπους περιφέρειες. Και αυτό το κάνουμε ακριβώς οι αντιπροσωπείες μας. Εμείς έχουμε και ένα δικό μας πρόγραμμα επικοινωνίας και ενημέρωσης για τα Δυτικά Βαλκάνια, το οποίο παρέχει σε αυτές τις αντιπροσωπείες το απαραίτητη χρηματοδότηση έτσι ώστε να ασκούν τη δραστηριότητά τους. Η ελόγω χρηματοδότηση βασίζεται στα ετήσια σχέδια επικοινωνίας των επιμένων αντιπροσωπείων. Άρα λοιπόν λαμβάνουμε υπόψη μας εμείς αυτά τα, αυτό τον ετήσιο σχεδιασμό και διαπιστώνουμε κατά πόσο πράγματι αυτά τα ετήσια σχέδια ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες μας, με τα θεματικά μας ε, παιδεία και ότι ακριβώς περιορίζονται σε θεματικά παιδεία έτσι ώστε να μην έχουμε απλά αποσπασματική ενημέρωση σε ό,τι αφορά κάθε επιμέρους μικρό project. Άρα λοιπόν αυτά ε, μπορούν να κάνουν αντιπροσωπείσμα ουσιαστικά τα πάντα. Ό,τι του ζητήσετε σε επίπεδο επικοινωνία, μπορούν να προβούν σε ενημερωτικέ εκστρατείε σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα θεματικά πεδία, μπορούν να έρθουν σε επαφή με του περιφερειακού φορεί. Και βέβαια μπορούν και είναι σε θέση να διαχειρίζονται τα ενημερωτικά κέντρα ε, και στις έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, σε κάθε πρωτεύουσα. Αλλά όχι μόνο στις πρωτεύουσες, υπάρχουν και σε μικρότερες πόλεις κάποια ε, ενημερωτικά κέντρα, info points όπως λέγονται, δηλαδή σε επίπεδο ε, αρχών τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Όλα αυτά λοιπόν χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα επικοινωνίας και ενημέρωσης. Και στο πλαίσιο του ίδιου εργαλείου προσπαθούμε να ασκήσουμε την πολιτισμική διπλωματία, δηλαδή με τη διοργάνωση σχετικών γεγονότων και στο πλαίσιο αυτό τα ενημερωτικά κέντρα ακριβώς λειτουργούν ως ε, κέντρα υποδοχής για τέτοιου είδους ε, πολιτιστικά γεγονότα. Κάθε είδους. Ε, φυσικά κάθε αντιπροσωπεία έχει και το δικό της media outreach, δηλαδή την μονάδα σε ό,τι αφορά την επαφή και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχει δηλαδή και λογαριασμός Twitter, ο οποίος είναι είναι πολύ σημαντικό εργαλείο, ειδικότερα αλλά και το Facebook για παράδειγμα για την περισσότερη ενημέρωση και των δημοσιογράφων και του τύπου. Και από εκεί και μετά μπορούμε να κάνουμε και κάποιες πιο συγκεκριμένες φυγομετρήσει προκειμένου να αντιληφθούμε καλύτερα το τι σκέφτονται το κοινό μας, οι ομάδες στόχοι μας ε, και σε σχέση με τη χρηματοδότηση. Ένα τέταρτο σημείο που θα ήθελα να θίξω είναι ο ρόλος που μπορούν να παίξουν οι εθνικές αρχές, γιατί δεν είναι αρμοδιότητα μόνο των ευρωπαϊκών αρχών να ε, προβούν σε αυτή την ενημέρωση και οι ίδιες οι κρατικές αρχές θα πρέπει να το κάνουν. Αν επιθυμούν δηλαδή να προσχωρήσει η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προβαίνει στην αντίστοιχη ενημέρωση του κοινού σε ό,τι αφορά τα όσα κάνει εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, πέρυσι διοργανώθηκε ένα σεμινάριο στο οποίο προσήλθαν και συνάδελφοι από τις διάφορες αντιπροσωπείες και από όλες τις ε, υπηρεσίες ε, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ολοκλήρωση ε, προκειμένου να συζητηθεί το ζήτημα της επικοινωνίας. Και πρόσφατα είχαμε και κάποιους πρέσβεις και προξένους προκειμένου να συζητήσουμε σημαντικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αυξηθούν σε επίπεδο επικοινωνίας. Και στο Μαυροβούνιο και τη Σερβία έχουμε ζητήσει την ενίσχυση των δυνατοτήτων που έχουν οι κρατικές αρχές προκειμένου να εφαρμόζουν τις σχετικές στρατηγικές ε, επικοινωνίε. Γιατί αυτό που συμβαίνει σε πολλέ περιοχέ είναι το να υπάρχει μια τέτοια στρατηγική ενημέρωση, αλλά να μην εφαρμόζεται λόγω έλλειψη των καταλήλων πόρων. Ένα πέμπτο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να θέξω, έξι σημαντικά είναι, οπότε ολοκληρώνω σιγά σιγά, ε, είναι το ζήτημα ε, τη στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια. Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική ανακοίνωση που παρουσίασε αυτή τη στρατηγική και πραγματικά βρίσκεται στο δημόσιο χώρο και γι' αυτό θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το έναυσμα που έδωσε η δημοσίευση αυτής στρατηγικής έτσι ώστε να τεθεί επιτάπητος για, τα για τους ενδιαφερόμενους φορείς αλλά και μέσω και μακροπρόθεσμα να ξεκινήσει μια ευρύτερη ένα ευρύτερο δημόσιο ε, διάλογο. Γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχει κάποιο σκεπτικισμό σε ό,τι αφορά περαιτέρω διεύρυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα πρέπει ε, στο πλαίσιο και των ε, της έναρξης των διαπραγματεύσεων να να ε, κάνουμε και τα όσα λέμε ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε. Άρα λοιπόν αυτή η δημοσίευση, η ανακοίνωση μάλλον τη στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια αποτέλεσε το έναυσμα για να ξεκινήσουμε μια ολόκληρη εκστρατεία ενημέρωση. Και για την ίδια τη στρατηγική δημιουργήσαμε μια ολόκληρη δέσμη ενημερωτικού υλικού, δηλαδή έχουμε fact sheets, εδώ διάφορα ενημερωτικά γραφήματα, ε, ενημερωτικά φυλάδια για κάθε μία επιμέρου χώρα. Ε, και εδώ προετοίμασα για εσά, Πρόεδρε, και ένα τέτοιο σετ από το έντυπο υλικό που έχουμε, αλλά από εκεί και μετά υπάρχουν και οπτικοακουστικά μέσα, για παράδειγμα βίντεο ε, σε ό,τι αφορά που παρουσιάζουν και ούχους, για παράδειγμα, οι οποίοι έχουν υποφεληθεί από αυτήν την προενταξιακή χρηματοδότηση. Έχουμε και κάποια information που ακριβώς ε, ε, διαφημίζουν το γιατί είναι ε, χρήσιμο για τη χώρα να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης εξηγούμε το τι ακριβώς είναι η διαδικασία της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι σημαίνει κράτη δικαίου, τι σημαίνει οικονομική διακυβέρνηση. Άρα λοιπόν εστιάζουμε σε αυτό το ενημερωτικό υλικό σε 4-5 σημαντικά σημεία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ειδικότερα σε ό,τι αφορά του διάβλου των μέσω ενημέρωσης. Όλα αυτά τα ε, υλικά είναι διαθέσιμα σε όλες τις ε, ε, χώρες των κρατών μελών της Ένωσης και κάποια έχουν μεταφραστεί στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Και φυσικά οποιοδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό το υλικό και να το εκτυπώσει έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσει στο πλαίσιο για παράδειγμα των δικών του παρουσιάσεων σε ό,τι αφορά τη δουλειά που κάνουμε στα Δυτικά Βαλκάνια. Και επίσης σε ό,τι αφορά την ενημερωτική εξαρτία που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαμε 8.000 ε, ε, προβολές ε, στο facebook, 5.000 στο twitter και 250.000 στο instagram και αυτό μόνο μέσα σε δύο ημέρες μιας παρουσίασης που κάναμε. Οπότε ε, όποιος παρακολουθεί τις δημοσίευσεις της Engineer μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες αυτές τις δημοσίευσεις. Και το έκτο σημείο τώρα είναι το τι θα ακολουθήσει στο άμεσο μέλλον. Υπάρχουν δύο ορόσημα, θέλετε, δύο σημαντικά σημεία σε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Ε, θα ξεκινήσει η ενημέρωση με το πρώτο πακέτο πρωταξιακή βοήθεια την διάσκεψη κορυφή ε, στη Σόφια ε, και την διάσκεψη του Ιουλίου. Εκεί θα χρειαστεί λοιπόν να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τι δικέ μα ομάδε ενημέρωση. Αλλά εκείνο που είναι ακόμα πιο σημαντικό και το κάνουμε ούτω ή άλλω είναι η όθηση που έχει δοθεί σε αυτή την ατζέντα να συνεχιστεί και στο ενδιάμεσο διάστημα. Ανάμεσα δηλαδή σε αυτά τα σημαντικά ορόσημα, έτσι ώστε να μην χαθεί ακριβώς αυτό το, αυτή η όθηση, όταν δεν υπάρχει κάποια ε, εκδήλωση υψηλού επίπεδου. Τι κάνουμε λοιπόν για να το επιτύχουμε. Δημιουργούμε μια σειρά από ε, διοργανώσεις ε, με, τις, ε, με την ακαδημαϊκή κοινότητα και με think tanks και στις ίδιες αυτές χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου ακριβώ να αυξηθεί και πάλι το ενδιαφέρον τη ακαδημαϊκή κοινότητα και το Think Tank για τα Δυτικά Βαλκάνια. Ήδη έχουμε προβλέψει κάποια events, ε, αλλά ε, ερχόμαστε σε επαφή ένεργα με τα think tank και τα, ε, πανεπιστήμια σε αυτές τις χώρες. Για παράδειγμα, πριν από δύο εβδομάδες διοργανώσαμε ένα τέτοιο, μια τέτοια μεγάλη εκδήλωση με έξι πανεπιστήμια από τα έξι διαφορετικά τις έξι διαφορετικές χώρες Δυτικών και από εκεί και μετά θα υπάρξει και ένα γεγονός όπου θα συμμετάσχουν και ε, δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι των ε, μέσων ενημέρωση που θα συναντηθούν με πολιτικού και εκπροσώπους τη Οργανωμένη κοινωνία των πολιτών προκειμένου να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση σε ό,τι αφορά και τη χρηματοδότηση, την προενταξιακή αλλά και την κατάσταση που ισχύει στι χώρε. Γιατί θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Δεν μπορούμε να θεωρούμε ω δεδομένο ότι γνωρίζουν ε, όλοι οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση το τι συμβαίνει στο επίπεδο τη προενταξιακή βοήθεια και το, και το ποια είναι η κατάσταση σε αυτέ τι χώρε των Δυτικών Αλβανίων. Άρα λοιπόν αυτό μπορεί να αποτελέσει μια καλή ευκαιρία προκειμένου να βρίσκεται στην ατζέντα μας η ε, η των Δυτικών Βαλκανίων. Επίση, συνεχίζουμε τη συνεργασία μα με του επαγγελματίε από το χώρο των μέσων ενημέρωση ε, και μετά από το αίτημα του Επιτρόπου Χάν, είχαμε και την ε, ε, η μέρα για τα μίντια, όπου στο πλαίσιο της οποίας 250 δημοσιογράφες εξέτασαν τα ζητήματα οικονομικής ανάπτυξης των δικών Αλβανίων, αλλά και της εκπαίδευσης, του επαγγελματισμού, του εγγραμματισμού, του ε, ε, ψηφιακού εγγραμματισμού των νέων και ούτω καθεξής. Αυτά τα ζητήματα θα εξεταστούν και πάλι στα επόμενα Media Days που έχουν προβλεφθεί για τους στην Σόφια και εκεί θα εστιάσουμε ιδιαίτερα και στους νέους δημοσιογράφους και πώς μπορούμε να τους υποστηρίξουμε. Επίση, προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε πιο στενά με τη Γενική Διεύθυνση επικοινωνία, την DG Computation, και θα προετοιμάσουμε ειδικότερα ε, πακέτα ενημερωτικά τα οποία ε, θα μπορεί και εκείνη η Γενική Διεύθυνση να χρησιμοποιεί στο πλαίσιο ε, της επαφή με τι δικέ τη ομάδε στόχους. Και από εκεί και μετά θα συνεχίσουμε προ ολοταχώ αυτή την περαιτέρω παρουσίαση τη σταθερικής για τα Δυτικά Βαλκάνια, διαχειριζόμενη όμω και τι σχετικέ προσδοκίε. Γιατί βέβαια δημιουργεί αυτή η στρατηγική μια σειρά από προσδοκίε, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να περάσουμε το μήνυμα ότι πολλά ακόμα θα πρέπει να γίνουν. Εδώ μιλάμε για το βέλτιστο δυνατό σενάριο, οπότε θα πρέπει πολλά να κάνουν αυτέ οι χώρε από την πλευρά του για να τα επιτύχουν όλα αυτά. Και έχουμε προβλέψει και ενημερωτικά σεμινάρια προκειμένου να εκπαιδευτούν όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτόν τον ε, τομέα, για παράδειγμα και το προσωπικό το οποίο είναι αρμόδιο για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων, προκειμένου να αντιλαμβάνεται ότι αυτά τα προγράμματα πράγματι θα πρέπει να έχουν μια σαφώ ορατή ευρωπαϊκή ταυτότητα, όπω αναφέρθηκε και από τον Επίτροπο πρόσφατα. Δηλαδή, από τον ίδιο το χαρακτήρα του τα προγράμματα θα πρέπει να είναι ταυτοποιήσιμα ω ευρωπαϊκά και σε ό,τι αφορά και τον αντίκτυπο που έχουν ε, στι ε, χώρε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι κρατικέ αρχέ των κρατών μελών, ε, έχουμε αξιοποιήσει ένα ε, πρόγραμμα αντίστοιχο του ΤΑΙΚΣ έτσι ώστε να υπάρξει μια αντιστοίχηση των επαγγελματιών αυτών των χωρών με επαγγελματίε από τι ε, από τις χώρες των κρατών μελών, ειδικότερα τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία προσχώρησαν τα τελευταία 15 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο υπάρχει δυνατότητα μεταβίβαση κάποιων επαγγελματικών δεξιοτήτων αυτών των εμπειρογνωμών στου επαγγελματίε των χώρων των Δυτικών Βαλκανίων και από εκεί και μετά υπάρχει ένα πρόγραμμα επικοινωνία outreach το οποίο θα ξεκινήσει του χρόνου ελπίζουμε και θα τρέξει για δύο-τρία χρόνια, ούτως ώστε να παίξει συμπληρωματικό χαρακτήρα προς τα όσα κάνουν οι αντιπροσωπείες, αλλά εστιάζοντας περισσότερο στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να κάνουμε και περισσότερες, ε, για παράδειγμα, ε, σφιγμομετρήσεις, ε, κατάρτιση επαγγελματιών και ούτω καθεξής. Αυτή λοιπόν η συνεργασία και με την Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας θα συνεχίσει στενά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα η Ρόζα Μπάλφουρ από το γερμανικό Marshall Fund των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ σήμερα. Ε, το πρώτο που πρέπει να πω είναι ότι η νέα στρατηγική της Γενικής Διεύθυνσης ΝΙΕΡ και της Περισσέξης Εξωτερικής Δράσης είναι η σωστή στρατηγική, πάει προς τη σωστή κατεύθυνση και δεν έχω σε καμία περίπτωση εδώ τη διάθεση να επικρίνω αυτή τη στρατική. Θα προσθέσω μόνο κάποια στοιχεία τα οποία ενδεχομένω να είναι χρήσιμα. Το πρώτο αφορά την κοινή γνώμη ε, στα Βαλκάνια. Ξέρω ότι υπάρχει ένα βαρόμετρο στα Βαλκάνια που λειτουργεί εδώ και 3-4 χρόνια χάρη στην, στο Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας και έρχεται να καλύψει ένα κενό. Ε, δείχνει πώς οι πολίτες στα Βαλκάνια βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Κωσφοπαίδιο, στην Αλβανία έχουμε πολύ υψηλά, υψηλές θετικές γνώμες. Στην υπόλοιπη περιοχή δεν είναι όμως το ίδιο και η πιο δύσκολη περίπτωση βεβαίως είναι η Σερβία. Ε, τα στοιχεία αυτά τα γνωρίζετε φαντάζομαι, αλλά αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ακόμα και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια σχετικά ε, φτωχή εικόνα, μια αρνητική εικόνα, πιστεύω ότι κυρίως είναι άγνωστη. Δηλαδή υπάρχει πολλοί που δεν γνωρίζει. Υπάρχει άρα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Ε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει κόσμος που έχει αρνητική ε, άποψη. Το θέμα είναι αυτοί που δεν γνωρίζουν αυτοί που, δεν, που θα πρέπει να αποτελέσουν το, στόχο της πολιτικής ε, επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντα σε ό,τι αφορά τους δείκτες για την κοινή γνώμη, ακόμα και αν γενικά τα στοιχεία δεν είναι και τόσο καθυσυχαστικά, όταν θέτουμε ερωτήματα συγκεκριμένα υλικά, υλική προτίμησης, οι πολίτες των Βαλκανίων κοιτάζουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, όταν είναι να ταξιδέψουν, όταν να εκπαιδευτούν, όταν είναι να βρουν δουλειά. Ε, σε υλικό επίπεδο λοιπόν, ακόμα και αν υπάρχει βεβαίως ανταγωνισμός και από άλλες ε, πλευρές και ακόμα και αν η Ρωσία ε, έχει γενικά μια πολύ θετική εικόνα στην περιοχή, όταν μιλάμε όμως για το υλικό σκέλος, κοιτάζουν οι πολίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι άλλη μια ευκαιρία λοιπόν για την πολιτική επικοινωνία της Ένωσης. Για τη Ρωσία τώρα και την παραπληροφόρηση έχουν εκφραστεί πολλές ε, ανησυχίες για το θέμα αυτό πρόσφατα και όλο και πιο πολλές εκθέσεις ε, προκύπτουν για το εύρος και το επίπεδο της ε, πολιτικής παραπληροφόρησης από τη Ρωσία στη Βαλκάνια. Εγώ θέλω να πω ότι ναι, βεβαίως συμβαίνει αυτό. Υπάρχει το Russia Today, Today το Serbia Sputnik, χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία έτσι ώστε να παίρνουν κάποια μηνύματα. Δεν είναι όμως η μόνη πηγή παραπληροφόρησης, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Η Τουρκία, οι χώρες του κόλπου, η Αλτζαζίρα, η Κίνα. Επίσης υπάρχουν εκπρόσωποι οι οποίοι παράγουν ε, παραπληροφόρηση και εκπρόσωποι εκπροσώπων σε τοπικό επίπεδο. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι βεβαίως πρέπει να μας ανισχύει το θέμα της παραπληροφόρησης αλλά θα πρέπει να το εντάξουμε στο πλαίσιό του δεν αφορά τη Ρωσία και το Κρεμλίνο που ε, χρηματοδοτεί την παραπληροφόρηση. Είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει στη Δυτικά Βαλκάνια όπως συμβαίνει και αλλού. Είναι σημαντικό να το εντάξουμε δηλαδή αυτό στο ευρύτερο πλαίσιο, να μην επικεντρωθούμε, να μην, να αποκλειστικά στην ρωσική παραπληροφόρηση. Στα Βαλκάνια βεβαίω είναι σημαντικό αυτό, διότι η Ρωσία έχει δεσμού ιστορικού με πολλέ χώρε. για να μπορέσει κανείς ε, να αντιμετωπίσει αυτή την παραπληροφόρηση με επίση ε, ακραίο τρόπο, αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη πόλωση. Πάντα η Ρωσία θα έχει θετική εικόνα σε αυτές τις χώρες, ό,τι και να γίνει. Οπότε, αντί να σχεδιάσουμε στρατηγικές ε, για να καταπολεμήσουμε την παραπληροφόρηση από τη Ρωσία, από τη Ρωσία ε, θα ήταν πιο σωστό να στέλνουμε ένα θετικό μήνυμα, ένα εναλλακτικό μήνυμα και μερικά ακόμα πράγματα ε, τα οποία θέλω να πω για το πώς ε, να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Ε, να σας πω ότι βεβαίως ότι από το 2014 και μετά η Ρωσία σίγουρα έχει αυξήσει την ε, καμπάνια παραπληροφόρησης ε, στην περιοχή για τους γνωστούς λόγους, για να υπονομεύσει η δηλαδή, τη Δύση, να την διαιρέσει. Η νέα στρατηγική της Ένωσης ε, για τη διεύρυνση είναι ένα πολύ θετικό βήμα προς σωστή κατεύθυνση και όλα όσα ελέγχθησαν την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και επικοινωνική διεύθυνση ΝΙΕΡ είναι επίση θετικά. Αυτό που θέλω να πω εγώ, που θέλω να προσθέσω, είναι 4-5 σημεία. Θα τα αναφέρω εν συντομία. Πρώτα απ' όλα να πιστεύω την προσοχή σας ε, για όσους ε, δεν το αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει μια έκθεση τη ομάδα ψηλού επίπεδου για τα fake news ε, και την επιγραμμική παραπληροφόρηση πρόσφατη έκθεση η γενική αρχή, οι γενικές αρχές νομίζω που αναφέρονται εκεί θα πρέπει να τις ασπαστούμε παντού στον κόσμο. Το βασικό είναι ότι χρειαζόμαστε μια ε, πολυδιάστατη προσέγγιση σε ό,τι αφορά την παραπληροφόρηση. Αυτή είναι ε, η σφαιρική προσέγγιση στην οποία αναφερθήκατε κι εσείς. Να πω επίσης, επίσης ότι είναι σημαντικό ε, ε, να συνδέσουμε τις προσπάθειες που γίνονται στα, πλαίσια της διεύρυνσης ε, με τις προσπάθειες που γίνονται στο εσωτερικό της Ένωσης. Δεν υπάρχουν χώρες που είναι πιο ευάλωτες από άλλες στην παραπληροφόρηση. Ε, Επίση πρέπει να συμμεριζόμαστε αυτές τις γενικές αρχές, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτές οι γενικές αρχές εφαρμόζονται και σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή σε το να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση σε τοπικό επίπεδο έχει σημασία να προσαρμοζόμαστε, να μεταφράζουμε, να προσαρμοζόμαστε στις τοπικές ε, ε, συνθήκες. Ε, να προσθέσω ότι δεν είναι μόνο θέμα επικοινωνίας και σχεδιασμού κάποιων εκστρατιών επικοινωνίας. Νομίζω ότι είναι εξίσου σημαντικό να καταρτίζουμε και αξιωματούχους που να μπορούν να συμμετέχουν σε συζητήσεις στην περιοχή, σε debate. Όχι να συζητάμε μόνο για τη διεύρυνση, να συζητάμε και τη δημόσια πολιτική γενικότερα. Ιδιαίτερα ε, σε ό,τι αφορά ζητήματα που έχουν, που έχουν σημασία για τους πολίτες της περιοχής. Για την υγεία, παραδείγματος χάρη τι σημαίνει μια πολιτική δημόσια υγεία που ανταποκρίνεται στι ανάγκε των πολιτών, Τι σημαίνει να έχουμε μια πολιτική εκπαίδευση που να αποτυπώνει τι ανάγκε ε, τη περιοχή και να έχουμε αξιωματούχου που να συμμετέχουν άμεσα στι συζητήσει αυτέ σε τοπικό επίπεδο. Δεν είναι μόνο θέμα πολιτική επικοινωνία, να συμμετέχουν άμεσα. Είναι ένα τρόπο ε, ε, να μην μιλάμε έτσι απλά για επικοινωνία γενικά, αλλά να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο. Ε, επίσης ζητήματα διαφάνειας, ζητήματα διαφθοράς, όχι μόνο ως μια συνθήκη, ε, μια προϋπόθεση για την ένταξη, αλλά ως ε, κάτι που είναι σημαντικό, ως ένα δημόσιο αγαθό. Ε, σε ό,τι αφορά τα μίντια, χρειάζεται μια προσπάθεια ε, μιλήσαμε για τα Media Days. Ε, αυτά έρχονται τώρα μετά από μια περίοδο ε, όμως που είχαμε, είχαμε ξεχάσει τα Βαλκάνια και έκτοτε τα πράγματα έχουν επιδεινωθεί. Η επικοινωνία του προηγούμενου μήνα ε, για πρώτη φορά ε, αναφέρει ότι το κράτος ε, ελέγχει υπερβολικά σε δυσανάλογο βαθμό τη ροή πληροφοριών και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί αυτό. Αυτό είναι κάτι που αναφέρεται και στην ομάδα υψηλού επίπεδου των εμπειρογνωμόνων. Το καλύτερο είναι να συνεργαζόμαστε με τα μίδια, να στοχοποιούμε μίδια ε, να αναπτύσσουμε στρατηγικές που να έχουν νόημα σε τοπικό επίπεδο και στα Βαλκάνια η κάθε χώρα έχει τις δικές της προκλήσεις σε ό,τι αφορά τα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχει ένα αίτημα από μελέτες, από έρευνες ε, για τα μέσα στα Βαλκάνια. Υπάρχει ένα αίτημα για κατάρτιση στην περιοχή, ε, ε, να υπάρχει μια ανθεκτικότητα των μίντια, να υπάρχει ηθική δημοσιογραφία, ερευνητική δημοσιογραφία. Πρέπει να βοηθήσουμε και τα μικρά τα μικρά μίντια να προστατευτούν από κυβερνοεπιθέσει, παραδείγματο χάρη, ε, θα ήταν καλό να υπάρξει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και τέτοιου είδου ε, βελτιώσει σε επίπεδο υποδομών. Πέρα από τα μίντια, πέρα από τα μέσα ενημέρωση, θα ήθελα να αναφερθώ στην ανάγκη συμμετοχή κοινωνία των πολιτών. Υπάρχει ένα project που αφορά την ε, ε, στήριξη κοινωνία των πολιτών από τι ΗΠΑ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω εδώ κάποια έγγραφα. Η Σερβία ήταν μία από τι χώρε τι οποίε εστιάσαμε στα Βαλκάνια. Έχουν λάβει χώρε σημαντικέ αλλαγέ ε, σε ό,τι αφορά το πώ προετοιμάζει τι υποστήριξει τη κοινωνία των πολιτών η Ευρωπαϊκή Ένωση στι διάφορε χώρε. Και ένα ζήτημα το οποίο έχει εξεταστεί και πρέπει να συνεχίσουμε να το εξετάζουμε είναι πώς ε, ε, θα μπορέσουμε να εμπλέξουμε ευρύτερα ένα ευρύτερο πεδίο κοινωνία των πολιτών, να μην επικεντρωνόμαστε λες στις πρωτεύουσες, ε, ε όχι δηλαδή η κοινωνία των πολιτών που ακολουθεί ήδη το δυτικό μοντέλο, που είναι ε, μορφωμένη, που είναι, μιλάνε πολλές γλώσσες. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και στην Ήπεθρο, να δούμε τι γίνεται στις τοπικές κοινωνίες, ίσως είναι ο πιο σημαντικός τρόπος ε, για να μπορέσουμε μέσω αυτών των τοπικών ε, debate, συζητήσεων, να έρθουμε σε επαφή με τους ε, πολίτες εκεί. Εάν γίνει αυτό στην Ήπεθρο, της στις θα πρέπει βεβαίω να διπλασιάσουμε το, το προσωπικό μας εκεί. Είναι σημαντικό λοιπόν να εντοπίσουμε τοπικούς παράγοντες να μπορούν να βοηθήσουν. Θα πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό στην πράξη βέβαια. Ο λόγος για τον οποίο δίνω έμφαση στους τοπικούς συνομιλητές είναι ότι έχουμε στοιχεία, έχουμε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ευρήματα για τη Σερβία, όπου έχουν γίνει πολλές μελέτες. Φαίνεται λοιπόν ότι ο τρόπος με τον οποίο οι ειδήσει επηρεάζουν τους πολίτες γίνεται μέσω ε, μιας φούσκας που δημιουργείται. Ε, το θέμα είναι να φτάσει κανείς σε αυτή τη φούσκα για να μπορέσει να επηρεάσει την πληροφορία και ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι μέσω των ανθρώπων. Ε, υπάρχουν επίσης στοιχεία ότι λιγότεροι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στις ειδήσει μέσω των μέσων ενημέρωσης, αλλά πιο πολύ τα μαθαίνουν από τους συγγενείς τους, τους φίλους τους. Πρέπει να βρούμε δηλαδή αυτές τις, ε, αυτούς τους κύκλους και να μπορούμε να μπορούμε να εμπλακούμε στις συζητήσεις εκεί. Αυτό βεβαίω ε, ε, εδώ λοχεύουν και κάποιοι κίνδυνοι, διότι όταν θα πρέπει να μιλήσουμε με ανθρώπου με του οποίου διαφωνούμε, να βρεθούμε σε δύσκολε συζητήσει. Και εδώ επανέρχομαι στο θέμα τη κατάρτιση. Γι' αυτό οι αξιωματούχοι θα πρέπει να είναι καταρτισμένοι για να μπορούν να αναλάβουν αυτά τα καθήκοντα που είναι κάπως πιο έτσι, απαιτητικά. Αυτά είχα να πω. Είμαι έτοιμος να, να ακούσω τι ερωτήσει σα. Έχω και το έγγραφο για την υποστήριξη τη κοινωνίας των πολιτών για όποιον ενδιαφέρεται. Ευχαριστούμε, αξιότιμη κυρία. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και ανοίγουμε τώρα τη συζήτηση. Επιτρέψτε, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω εγώ ως εισηγήτρια για τις στρατηγικές επικοινωνίες. Θα αλλάξω λίγο τη μέθοδο που χρησιμοποιώ στις συζητήσεις αυτής της Επιτροπής. Να αναφερθώ πρώτα στα όσα παρουσίασε μόλις η κυρία Μπαλφόρ. Έχετε δίκιο. Δεν εστιαζόμαστε εδώ μόνο στη ρωσική προπαγάνδα. Δεν λέγεται κάτι τέτοιο στην έκθεση της οποίας εισηγήτρια ήμουν εγώ και εκεί παρουσιάζουμε το γεγονός ότι υπάρχει και προπαγάνδα ε, που ουσιαστικά δεν έχει κρατικό χαρακτήρα όλη αυτή η προπαγάνδα που παρουσιάζεται στον Νότο και από άλλα κράτη μάλιστα αλλά ήθελα να πω ότι πραγματικά τα Δυτικά Βαλκάνια είναι η παιδική χαρά του Θεού ε, ε, ονόμαζαν έτσι την Πολωνία παλιά. Είναι μια παιδική χαρά, ένα χωνευτήρι πολλών επιρροών. Γιατί εστιαζόμαστε σε αυτό, στις αλλαγές μοτίβων ε, ρωσικής προπαγάνδας, ε, ειδικότερα το 2014 και μετά. Πρώτα απ' όλα, μας απασχολεί η εγκύτητα της περιοχής. Το ίδιο συνέβαινε και στην Ουκρανία. Ε, που επίση επηρεάζει και τα Δυτικά Βαλκάνια και είναι σαφέ ότι εντάθηκαν οι δραστηριότητε εκείνη την περίοδο, αλλά υπάρχει και ένα επιπλέον παράγων. Πιστεύω πολύ σημαντικό για τα Δυτικά Βαλκάνια αλλά όχι μόνο ε, στα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά και στην Γεωργία και αλλού. Στην αρχή αυτής της θητείας ε, της ε, Κομισιόν και του Κοινοβουλίου, δεν υπήρχαν προοπτικές για το μέλλον, ούτε προοπτικές διεύρυνσης στο προβλέψιμο μέλλον. Και αυτό ήταν θλιβερό για αυτές τις κοινωνίες. Ευτυχώς το τελικό αποτέλεσμα είναι πάνω από θετικό. Οπότε αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε αυτή τη στρατηγική κατά αυτής της αίσθησης κόπωσης, δυσαρέσκειας, έλλειψης ε, ελπίδας ε, στις περιοχές αυτές. Έτσι ενισχύσαμε λοιπόν τις ε, δράσεις μας, ε, κάτι που θεωρώ ότι παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία ε, και μεταξύ των θεσμικών συνομιλητών μας, διότι αναλύθηκαν δράσεις που ήταν απαραίτητες φυσικά και εδώ είναι η ερώτησή προς τους δύο κυρίους Πώς προτίθεστε να προσεγγίσετε αυτό το διτό φαινόμενο με το ρωσικό φυσικά και τα άλλα που ακούσαμε στις προηγούμενες παρουσιάσεις. Δηλαδή, ε, ποιες πρακτικές δράσεις θα αναλυθούν από τα θεσμικά όργανα. Θα εστιαστούμε στην πρόληψη και καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, ε, στην καταπολέμηση της επιρροής των ριζοσπαστικών οργανισμών και ιδεολογιών, Αλλά παρόλα αυτά σε αυτές τις στρατηγικές επικοινωνίες θα πρέπει να κάνουμε και άλλες παράλληλες προσπάθειες. Αλλά έχετε δίκιο, αξιότιμη κυρία, με αυτούς τους κλειστούς κύκλους, αυτές τις φούσκες ενημέρωσης, ε, θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Πιστεύω ότι αυτές οι φούσκες, αυτοί οι περιορισμένοι κύκλοι, όπου κυκλοφορούν συγκεκριμένες πληροφορίες, σχετίζονται ακριβώς με αυτή την δυσαρέσκεια, την απελπισία που είδαμε παλιότερα. Γιατί τώρα παρατηρούμε ότι τόσοι πολλοί οργανισμοί και θεσμοί κάνουν τόσε πολλέ προσπάθειες που κατά την άποψή μου έχουμε φτάσει ε, έχουμε αποκτήσει την απαραίτητη ορμή. Όπως βλέπετε, ακούμε πολύ ενδιαφέρουσες φωνές, έχουμε εκπροσώπους ε, της Ανεξάρτητης Ένωσης Δημοσιογράφων της Σερβίας ε, εδώ μας επισκέπτονται νομίζω μάλιστα με χορηγία από κάποιον από την Τιτζινίαρ μάλλον η κυρία Βάζιτς Νίκολιτς έχετε το λόγο έχουμε περιορισμένο χρόνο οπότε παρακαλώ να είστε σύντομοι ευχαριστώ Καλημέρα. Λέγομαι κύριε Βάση Νικολίτσα από τον Ανεξάρτητη Ένωση Δημοσιογράφων τη Σερβίας. Με συνοδεύουν οι συνάδελφοι από το Μαυροβούνιο, ο Ράνταμιν Κράσκοβιτ, αντιπρόεδρο των συνδικάτων των δημοσιογράφων του Μαυροβουνίου και ο συνάδελφος εδώ από την Ένωση Δημοσιογράφων τη Φύρωμα και από την Ένωση Δημοσιογράφων η συνάδελφο μου από εδώ, από τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Καλύπτουμε ουσιαστικά όλους τους δημοσιογράφου των Δυτικών Βαλκανίων. Μας ζήτησαν να σχολιάσουμε κάποια τα ζητήματα εδώ εγώ. Να σας πω ότι επιδοκιμάζουμε την ιδέα της στρατηγικής επικοινωνίας. Διότι στη Σερβία και γενικότερα στα Δυτικά Βαλκάνια τα αποτελέσματα των προγραμμάτων και των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι τόσο ορατά όσο θα έπρεπε. Πολλές έρευνες μάλιστα δείχνουν ότι στη Νότια Σερβία θεωρείται η Ρωσία ως μεγαλύτερος χορηγός, ενώ δεν είναι, αν κοιτάξει κανείς τα νούμερα. Θα ήθελα επίσης να τονίσω όσον αφορά τις στρατηγικές επικοινωνίες πόσο σημαντικό είναι όταν εξωματούχοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχονται στη Σερβία να έρχονται σε επαφή όπως είπε η συνάδελφος ε, να έρχονται σε επαφή με τα μέσα με, τους, ε, με τις δημοσιογράφων με τα επαγγελματικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που τηρούν κάποια πρότυπα, διότι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είχαμε περιπτώσεις όπου δόθηκαν συνεντεύξεις στα μέσα που είναι γνωστά για την ανηθικότητά τους για τις ε, εκστρατείες λασπολογίας κατά δημοσιογράφων κτλ. Οπότε σκεφτείτε το και αυτό στο πλαίσιο των στρατηγικών επικοινωνιών, διότι ε, πρέπει να ακουστεί η φωνή σα ε, στους πολίτες οι οποίοι είναι υπέρ τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Αν πάτε στα άλλα μέσα, τότε αυτοί οι πολίτες οι πρώτοι αισθάνονται προδομένοι. Αναφέρατε και πολλά άλλα πράγματα για τα οποία θα ήθελα να πω κάτι. Να σας πω τι κάνουμε εμείς σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Για παράδειγμα, οι φούσκες αυτές που αναφέρθηκαν, οι κλειστοί κύκλοι, ε, ειδικότερα Σερβία, και πιθανότητα επαναλαμβάνω και στις υπόλοιπες περιοχές ε, οι πληροφορίες που περνούν στόμα με στόμα, οι φημολογίες. Γιατί συμβαίνει αυτό, πρέπει να αναρωτηθούμε, διότι η εμπιστοσύνη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, έχει υποβαθμιστεί. Οι άνθρωποι βασίζονται στους φίλους και γνωστούς τους. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της δεκαετίας του 90. Ξέρετε τι ρόλο έπαιξαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το η δεκαετία του 90, το γνωρίζουμε όλοι. Ε, σχετίζεται επίσης και με το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι δημοσιογράφοι και τα μέσα μαζική ενημέρωση στη Σερβία. Από αυτέ τι χώρε και λείπει το κοσφόπεδο τη σημερινή εκδήλωση. Έχουμε ένα κοινό πρόγραμμα. Δεν ήρθα να το διαφημίσω, μπορείτε να το δείτε στην εκθεσή μα. Προσπαθούμε μέσω αυτού του προγράμματο να εστιαστούμε στην νομική προστασία των μέσων μαζική ενημέρωση και στι ελευθερίε των δημοσιογράφων αλλά και στην ασφάλεια των δημοσιογράφων. Κάτι πολύ σημαντικό για την τελευταία διετία Είχαμε 434 σωματικές επιθέσεις, απειλές, ε, παρακολουθήσεις δημοσιογράφων. Συνήθως ε, δημοσιογράφων που επικρίνουν τις κυβερνήσεις. Οι δημοσιογράφοι μας λοιπόν εργάζονται σε δεινές ε, συνθήκες. Και φυσικά νομοθεσία υπάρχει, αλλά δεν υλοποιείται. Αυτό είναι σημαντικό γιατί μιλάμε για το περιβάλλον, το περιβάλλον μέσα στο οποίο εμείς θέλουμε να καταπολεμήσουμε την παραπληροφόρηση, τα fake news στην Σερβία. Τι ζούμε την παραπληροφόρηση. Ζούμε με αυτά. Οι πολίτες μας δεν ξέρουν όταν διαβάζουν οτιδήποτε αν είναι αληθές ή όχι. Και δυστυχώς πολύ περιεχόμενο εμφανίζεται σε ταμπλέτες ή στην τηλεόραση το οποίο δεν είναι πραγματική είδηση αλλά περισσότερο προπαγάνδα. Όλο αυτό είναι κομμάτι φυσιολογικό της ειδησιογραφίας της χώρας μας. όταν μιλάμε για fake news, για ψευδείς ειδήσει που επηρεάζονται από ξένες δυνάμεις όπως αναφέρατε, όχι μόνο έχουμε πρόβλημα με το να μάθουμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, από ποιον προέρχονται, ούτε καν ξέρουμε ποια είναι η χρηματική ροή. Τόσο από τους ξένους, αλλά και από τους συμμεδαπούς. Δεν ξέρουμε ποιος χρηματοδοτεί ποια μέσα, ποιος είναι ιδιοκτήτης ποιου μέσου. Το πρόβλημα λοιπόν είναι περίπλοκο και ξέρω ότι το γνωρίζετε όλοι σας. Αναφέρατε αυτές τις εκθέσεις ε, και τα λοιπά, αλλά είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι αν οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους χωρίς να φοβούνται για τη ζωή τους και την οικονομική τους ε, επιβίωση, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν το δημοσίο συμφέρον. Και αν δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, τότε οι πολίτες των χωρών αυτών δεν μπορούν να κάνουν επιλογές βάσει ενημέρωσης. Και αν δεν μπορούν να κάνουν τέτοιες επιλογές βάσει ενημέρωσης, έχουμε πρόβλημα που έχουμε ήδη ουσιαστικά. Αυτά προσπάθησα να είμαι σύντομη. Αν έχετε ερωτήσεις για μένα για τους συναδέλφους μου εδώ, παρακαλώ ενημερώστε μας. Μα ζητήσετε να πούμε κάτι για τη ρωσική επιρροή στα Δυτικά Βαλκάνια. Ε, Πρόεδρο, παρακαλώ, κλείστε, διότι πρέπει να δώσω το λόγο και στου βουλευτέ. Ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, θα έλεγα ότι το συμπέρασμα είναι πω ε, για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα, πρώτα Πρέπει να διασφαλίσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για τους δημοσιογράφους και τα μέσα. Να έχει αναπτυχθεί ένα επαρκώς ασφαλές περιβάλλον και να διασφαλίσετε η ύπαρξη του κράτους δικαίου σε αυτές τις χώρες. Αυτά. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρος. Ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ και που μας μιλήσατε. Να καλωσορίσω και τους υπόλοιπους δημοσιογράφους, ειδικότερα τον εκπρόσωπο από τη Βοσνία Ερσεγοβίνη. Θα πάμε στη χώρα σας αμέσως μετά το Πάσχα και το προηγούμενο σημείο της συζήτησής μας αφορούσε την κατάσταση ασφαλείας εκεί και τις δραστηριότητες της Eurofor ε, Αρθέα. Απλά ενημερωτικά σας το λέω. Ο κύριος Στέτινα θέλει να μιλήσει. Ωραία. Ο κύριος Πίτσουλα πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, να ευχαριστήσω και όλους τους ε, ομιλητές γιατί μας παρουσίασαν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το τι συμβαίνει και πώς αυτή η στρατηγική ε, διεύρυνση που περιμένουμε τόσο καιρό θα μπορέσει να λειτουργήσει στην πράξη. Είναι περιορισμένος ο χρόνος. Ε, τώρα εγώ είμαι από το πιο καινούριο κράτος μέλος της Ένωσης, στην Κροατία η ακόμα φρέσκες μνήμες ε, σε ό,τι αφορά προκλήσεις που χρειαστήκε να ξεπεράσουμε. Σε γενικές γραμμές, η διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δύσκολο να, την πουλήσει κανείς ε, στους πολίτες των κρατών μελών. Η προσχώρηση όμως ε, είναι όλο και πιο δύσκολη για, τους, για τα νέα μέλη. Νομίζω πως ήταν πολύ πιο απλό να δημιουργηθεί το 1957 η ΟΚ από το να προσχωρήσει κάποιος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 60 χρόνια μετά. Οπότε ε, ελπίζω αυτή η νέα στρατηγική να είναι αξιόπιστη ε, και να είναι και πραγματοποιήσιμη. Ακούγοντάς σας πολύ προσεκτικά, νομίζω ότι είναι σημαντικό η στρατηγική αυτή να προσαρμοστεί να δώσουμε μια αίσθηση οικειοποίηση σε τοπικό επίπεδο, διότι μιλάμε για διαφορετικές χώρες ε, στα Δυτικά Βαλκάνια και η στρατηγική αυτή γίνεται αντιληπτή διαφορετικά από την κάθε χώρα. Και στη Βοσνία έχουμε τρεις ομάδες διαφορετικές. Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Μακεδονία ε, Κόσοβο, Βοσνία, Τζεχοβίνη και κάτι άλλο που είναι σημαντικό με βάση τις εμπειρίες που έχουμε συλλέξει θα πρέπει να εντοπίσουμε τις ομάδες βέτο δηλαδή τις ομάδες εκείνες πολιτών που θέλουν οπωσδήποτε να περισπιστούν ένα status quo διότι τα συμφέροντά τους πλήττονται από τι μεταρρυθμίσει, Μιλάμε για ομάδε που έχουν επιρροή, όχι απαραίτητα πολιτικέ ομάδε ή πολιτικέ ελίτ. Παραδείγματο χάρη ε, οι βετεράνοι του πολέμου, ε, οι δημόσιοι υπάλληλοι, κάποιοι βιομήχανοι και βεβαίως ε, σημαντικοί επιχειρηματίες που έχουν έχουν επαφέ. Δεν συμμετέχουν σε εκλογές, αλλά επηρεάζουν εκλογέ. Θα πρέπει αυτέ τι ομάδες να τις εντοπίσουμε στην κάθε χώρα και να προσπαθήσουμε να πιέσουμε ε, προ του πολιτικού ηθήνοντε, του πολιτικού προ την σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ο Γιώζα Ράντο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του πάνελ για την εισαγωγή. Η στρατηγική επικοινωνίας ε, είναι αναπόσπαστο μέρος οποιασδήποτε διαδικασίας ένταξης, αλλά αυτές οι στρατηγικές έχουν αποτύχει στο να φτάσουν στον τελικό αποδέκτη, δηλαδή στους πολίτες της κάθε χώρας. Φτάνουν ε, στις πολιτικές ελίτ, στις κοινωνικές ελίτ, που ούτως ή άλλως ε, είναι γνωστές οι απόψεις τους, ε, είναι ενημερωμένοι ήδη. Και αυτό, δεν, και αυτό οι στρατηγικές οι δεν είναι, δεν είναι στρατηγικές αλλά υπάρχουν παράσιτα στο μήνυμα που προσπαθούμε να περάσουμε. Υπάρχουν εμπόδια και τα μέσα ενημέρωσης εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε αυτήν την, την στρατηγική. Η κατάσταση με τα μέσα ενημέρωσης, το περιβάλλον, το μηντιακό στις χώρες αυτές δεν έχει βελτιωθεί τα τελευταία 5-6 χρόνια. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση παρεμφερή, ε, το κράτος ε, ελέγχει τα μίντια, ε, δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες, ε, υπάρχει μια έτσι αδιαφάνεια, είναι χαμηλό το επίπεδο επαγγελματισμού, ε, υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα στο τεφό της εργασιακής σχέσης στα μέσα ενημέρωσης. Οι στόχοι λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να περιλαμβάνουν και τα μέσα ενημέρωσης. Όπως υπήρξε ξεχωριστή στρατηγική για το δικαστικό τομέα, με κοινού στόχου, με παράλληλη εποπτεία της διαδικασίας μεταρρύθμισης ε, ε, σε ό,τι αφορά τη δικαστική εξουσία. Κάτι αντίστοιχο ε, θα πρέπει να αποτελεί στόχο του σχεδίου δράσης για τον τύπο ή στα πλαίσια των έξι πρωτοβουλειών. Θα πρέπει να αφιερώσουμε μια ειδική στρατηγική για τα μέσα ενημέρωσης. Αν θέλουμε να πετάσουμε στους πολίτες δεν γίνεται χωρίς ελεύθερα και ε, αμερόληπτα μέσα ενημέρωσης. Οι δυσκολίες ε, είναι παρεμφερείς ε, με τις δυσκολίες στο δικαστικό τομέα. Θα πρέπει λοιπόν να το κάνουμε αυτό και για τα μέσα ενημέρωση. Δεν ξέρω αν η Κομισιόν σκοπεύει να κάνει κάτι τέτοιο και δεν ξέρω αν έχουν σχολιάσουν αυτή την πρόταση τα μέλη του πάνελ. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Έτιερ. Ευχαριστώ. Ακούσαμε πολλά και ενδιαφέροντα στις παρουσιάσεις. Από ό,τι φαίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει μεγάλη έμφαση στη στρατηγική επικοινωνίας, ιδιαίτερα στα Δυτικά Βαλκάνια. Πολλά χρήματα επενδύονται, όμως δεν ε, φέρνει αποτέλεσμα αυτή η προσπάθεια. Η κυρία Μπάλφορτ προηγουμένως αναφέρθηκε στις μελέτες της, στις μελέτες σύμφωνα με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καλή εικόνα εκεί. Και οι λόγοι γι' αυτό είναι ότι οι πολίτες δεν γνωρίζουν αρκετά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ μόνο μερικώς δεν νομίζω ότι μπορούμε να το γενικεύσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Παραδείγματο χάρη, στη Μακεδονία πριν από 10 χρόνια ήδη πληρούσαν όλε τι προϋποθέσεις για να ξεκινήσουν τι διαπραγματεύσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώ η χώρα αυτή είναι ακόμα στο, στα, στην αίθουσα αναμονής. Οι, οι πολίτες της Μακεδονίας ε, γνωρίζουν τη μήνυμα στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το μήνυμα αυτό δεν είναι θετικό, ούτε καλό. Πώς λοιπόν μπορείτε να ε, επαναφέρετε την εμπιστοσύνη των πολιτών της Μακεδονίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο μέτρα, δύο σταθμά. Ε, για να δούμε πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Χθες μίλησα με Μακεδόνες πολίτες οι οποίοι θεωρούν ότι υπάρχει πίεση αυτή τη στιγμή στη Μακεδονία να αλλάξει όνομα. Πράγματα που επηρεάζουν την ταυτότητα της χώρας και αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση σιωπά. λες και είναι ένα φυσιολογικό δρόμο για την προσχώρηση στην Ένωση. Μπορούν να εμπιστεύονται μια τέτοια πολιτική οι Μακεδόνες. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να αλλάξουμε την ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στα Δυτικά Βαλκάνια. Αυτό είναι το πρώτο. Και θα πρέπει να αλλάξουμε και την πολιτική απέναντι στη Μακεδονία έτσι ώστε να μπορεί να υπάρξει μια σωστή επικοινωνία και να γίνουν οι, οι πολιτικές μας κατανοητές προς τους πολίτες. Ευχαριστώ. Εάν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις από τους ευρωβουλευτές, να δώσω το λόγο ε, στους πανελίστες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για αυτά τα ερωτήματα. Θα είμαι πολύ σύντομο. Ε, γιατί γνωρίζω ότι έχουμε πλήρωση χρόνου. Θα ήθελα να επανέλθω σε τρία-τέσσερα σημεία που αναφέρθηκαν. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά το ζήτημα τη παραπληροφόρηση, συμφωνώ με τα όσα υπόθηκαν. Είναι πολύ περιπλοκό το ζήτημα και όπω ε, είπε και η Μπαρφούρτη, εγώ σα ε, συνιστώ να υπάρξει μια έκθεση από την ε, ψηλό επίπεδο ομάδα εμπειρογνωμόνων. Όπω γνωρίζετε, οι συνάδελφοι από την Επιτροπή ήδη προετοιμάζουν μια ανακοίνωση σε σχέση με αυτό το ζήτημα ε, και ε, δύο βασικέ κατευθύνσει θα ακολουθήσει αυτή η ανακοίνωση. Είναι καταρχήν η διαφάνεια ως προς το ποιο χρηματοδοτεί τι, ποια είναι η πηγή της κάθε πληροφορίας και ποια είναι η προηγούμενη πηγή από κάθε πηγή, για να αντιλαμβανόμαστε δηλαδή ε, ποια είναι η αλυσίδα αν θέλετε της ε, πληροφορίας. Και δεν θα αναφερθώ περαιτέρω σε αυτό. Υπάρχουν ε, εργασίες που συνεχίζονται από τη δική μας πλευρά και από την πλευρά της υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Θα αξιοποιήσουμε δηλαδή τις ενέργειε που έχουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άλλο ζήτημα των bubbles, ε, αυτές οι δηλαδή, ίσως ε, αποτελεί πραγματικά ένα μεγάλο, μια μεγάλη πρόκληση για όλους τους επαγγελματίες από το χώρο της ενημέρωσης. Ε, θεωρώ πως εδώ έχουμε να κάνουμε το πρόβλημα του εξαιρετικού κατακαιρματισμού του το κοινού μας, ακόμα και στις δικές μας χώρες, πράγμα το οποίο καθιστά πολύ δύσκολη την χάραξη γενικότερων ενημερωτικών στρατηγικών. Πράγμα το οποίο τελικά με φέρνει σε αυτό που ανέφεραν μία σειρά από ευρωβουλευτές, σε ό,τι αφορά δηλαδή ε, την παροχή ειδήσεων που είναι πολύ εξειδικευμένες και εξατομικευμένες σε ό,τι αφορά το κάθε κοινό. Εγώ ε, πιστεύω πάρα πολύ ε, στο να αλλάζουμε μία στρατηγική επικοινωνιακή. όχι δηλαδή ως προς το περιεχόμενο της ίδιας της ενημέρωσης, αλλά ως προς την προσαρμογή του περιεχομένου στο, στο, κοινό, δηλαδή το να βλέπουμε ποιο είναι το κοινό μας. Ένα ακόμα ζήτημα που αναφέρθηκε είναι αυτό το μέσο ενημέρωσης, στο media. Ε, το ανέφεραν ήδη οι συνάδελφοι, είναι κέρια σημασίας και ε, το παρακολουθούμε φυσικά από κοντά, ο Κλάου θα το αναφέρει, αποτελεί μία από τις ε, προτεραιότητε μας. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα το λόγο. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Σε ό,τι αφορά τα μέσα ενημέρωση, προφανώ εδώ η κατάσταση είναι ένα ζήτημα που ανησυχεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις ε, και αναφέρεται με ιδιαίτερη έμφαση αυτό το ζήτημα στις εκθέσεις μας, ε, στην έκθεση για παράδειγμα του Απριλίου θα δείτε ότι καλύπτουμε το ζήτημα της κατάστασης των μέσων ενημέρωση σε κάθε μία από αυτές τις χώρες και μάλιστα με αρκετό βαθμό λεπτομέρειας. Ε, παρακολουθήσαμε τις εξελίξεις επί σειρά ετών και ήδη έχουμε κάποιους δείκτες μέτρησης σε ό,τι αφορά τα μέσα ενημέρωσης Και δεν έχουμε μόνο τις αναφορές σε κάθε χώρα, αλλά έχουμε και ανταλλαγή απόψεων με τους ε, επαγγελματίε από το χώρο ε, της ε, ενημέρωσης. Για παράδειγμα, κάθε δεύτερο χρόνο διοργανώνουμε και μια σχετική διάσκεψη και τα όσα μαθαίνουμε στο πλαίσιο αυτών των διασκέψεων μας οδηγούν στο να διαπιστώνουμε το τι ακριβώς πρέπει να γίνει, τι καινούριο πρέπει να γίνει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε, αλλά και να χρηματοδοτήσουμε ενδεχομένως αλλά και να ενισχύσουμε την σχετική εμπειρογνωμοσύνη, για παράδειγμα και την δικαστική εμπειρογνωμοσύνη ε, σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης σε ό,τι αφορά την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθεροτυπία. Επίσης, εξετάζουμε και την αύξηση της αξιοπιστίας, την εμπιστοσύνη δηλαδή στα μέσα ενημέρωσης, τη δημιουργία για παράδειγμα μια νέα αρχής, αλλά και υποστήριξη σε ό,τι αφορά τα δίκτυα των δημοσιογράφων, αλλά και την παροχή εκπαίδευση. Όλα αυτά ως ιδέες προέκυψαν μετά ακριβώς τις συζητήσεις που κάνουμε κάθε φορά με τους εκπροσώπους αυτού του χώρου αλλά και τις οργανώσεις της ε, κοινωνίας των πολιτών. Και μετά από την τελευταία συνάντηση τον ε, Νοέμβριο του 2017 ε, συμφωνήσαμε με τη CBRD το να ε, δούμε κατά πόσο μπορούμε να ε, παράσχουμε και κάποια χρηματοδοτική υποστήριξη και στο Endowment for Democracy καθώς ε, μπορεί να βοηθήσει και μικρές και νεοφυείς επιχειρήσεις που χρειάζονται ακριβώ κάποιο αρχικό κεφάλαιο για να ξεκινήσουν τη λειτουργία του, χωρί να χρειάζεται εκεί να γίνει κάποιο, κάποιος κάποια ιδιαίτερη διαδικασία ε, προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντο. Ε, αυτό δηλαδή το endowment, ε, όπω κατέστησε σαφέ και στη διάσκεψη, είναι διαθέσιμο και υπάρχει κατάλληλη χρηματοδότηση την οποία παρέχει για τέτοιου είδου επιχειρήσει. Αυτή λοιπόν η χρηματοδοτική περίοδος 2014-2020 ε, ανέρχεται συνολικά σε 20 εκατομμύρια ευρώ για τα Δικά Βαλκάνια και την ε, ε, Τουρκία. Φυσικά δεν έχουμε μεγάλα ποσά χρηματοδότηση εδώ, αλλά ακριβώ επειδή έχουμε να κάνουμε μικρού φορεί, μικρά μεσανημερώσει, δεν χρειαζόμαστε για πάρα πολλά τέτοια κονδύλια. Και στην επόμενη διοργάνωση των Media Days στα Σκόπια, θα έχουμε τη δυνατότητα για μία ακόμα φορά να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. Σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα τώρα τη ε, ε, φούσκα του Bubble και όπω αναφέρθηκε και στο πλαίσιο τη συνάντηση τη ομάδα υψηλού επίπεδου εμπειρογνωμόνων, ε, είναι το ότι αυτά τα μέσα κοινωνική δικτύωση είναι τα λιγότερο αξιόπιστα ω πηγέ πληροφορία. Δηλαδή, ό,τι διαβάζει εκεί κανεί δεν θα πρέπει αυτομάτω να το εμπιστεύεται. Νομίζω πω η ομάδα υψηλού επίπεδου το ανέφερε αυτό με ξεκαθαρό ότι θα πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη μας ακόμα και στο πλαίσιο της επικοινωνίας που κάνουμε ακριβώς μέσω των μέσων ε, κοινωνικής δικτύωσης αφού και εμείς τα χρησιμοποιούμε για επικοινωνικούς σκοπούς. Ε, θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιου διάβολου ακολουθεί η επικοινωνία μας. Και από εκεί και μετά ε, θα πρέπει να δούμε, όπως είπε και ο Λούς στο πλαίσιο τη ομάδα του, με βάση την πολιτική που ακολουθούμε ποιε είναι οι ανάγκε της, ε, της κάθε ομάδα στόχου, του κάθε κοινού μα, έτσι ώστε να προσαρμόσουμε καλύτερα τι ε, πληροφορίε μα στι ανάγκε του. Ε. ε, όπως ανέφερε και ο κύριο Πίτσουλα, δηλαδή ε, αυτές τις ιδιαίτερες ομάδες στις οποίες θα πρέπει να κατευθύνουμε την ενημέρωσή μα. Και τέλο, σε ό,τι αφορά την πιο περιφερειακή προσέγγιση, δηλαδή σε περιφερειακό επίπεδο και τη χρήση κατά τόπους, κατά τόπους γλωσσών. Ναι, αναφέρθηκε αυτό και το γνωρίζουμε. Χρειαζόμαστε δηλαδή και περισσότερο προσωπικό, αλλά με τα ε, εφιστάμενα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μα προσπαθούμε να κινηθούμε και πέραν των πρωτεύουσων. Για παράδειγμα, η αντιπροσωπεία στη, στα Σκόπια έχει ξεκινήσει μια μεγάλη ενημερωτική εκστρατεία σε ό,τι αφορά περιβαλλοντικά ζητήματα. Δηλαδή ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι και τόσο αμφιλεγόμενο, δεν αφορά δηλαδή ανθρώπινα δικαιώματα ή του δικαίου αλλά το οποίο αναφέρεται ακριβώς στην προστασία του περιβάλλοντος και στο ότι αυτό αποτελεί όφελο για τους ανθρώπους. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της ενομερητικής εξαρτίας κατευθύνθηκαμε στις μικρότερες κοινότητε και τους Δήμους και είχαμε και τον ε, προσδευτή από την πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση με ε, πρέσβε από ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου ακριβώς να επισκεφτούν μικρούς Δήμους και κοινότητε, να επισκεφτούν τα έργα που λαμβάνουν χώρα εκεί και να προβούν σε αυτή την ενημέρωση. Αυτή λοιπόν η αξιολόγηση που έγινε σε συνέχεια αυτών των επισκέψεων ήταν πολύ θετική γιατί αυξήθηκε κατακόρυφα η ορατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και η κατανόηση ως προς τα περιφαλωτικά ζητήματα. Μια αντίστοιχη ενημερωτική εκστρατεία έλαβε χώρα στο Μαυροβούνιο ε, σε ό,τι αφορά την διαχείριση των αποβλήτων. Εάν ε, κανεί ε, δει για παράδειγμα τα Δυτικά Βαλκάνια του τι συμβαίνει στου δρόμου, θα διαπιστώσει ότι τα σκοπίδια αποτελούν ένα πρόβλημα. Και εκεί λοιπόν ε, με, χρησιμοποιήσαμε φημισμένους ε, αθλητές από τις ομάδες handball και μπάσκετ της χώρας οι οποίοι προσπάθησαν να εξηγήσουν ακριβώς το γιατί θα πρέπει να έχουμε μια διαφορετική ε, συμπεριφορά σε ό,τι αφορά τα απορρίμματά μας και πραγματικά καταφέραμε να φτάσουμε εδώ στο, στο μισό πληθυσμό του Μαυροβουνού. Μετά, στην Αλβανία είχαμε μια διαφορετική κατάσταση, αν θέλετε, ένα διαφορετικό πρόγραμμα όπου 40 με 50 δήμοι και κοινότητες ε, ε, εκδήλωσαν ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τη λήψη υποστήριξη αλλά και εκπαίδευση, σε ό,τι αφορά κάποια ε, focal points που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν, σε ό,τι αφορά ζητήματα Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία αφορούν ιδιαίτερα το κοινοτικό και περιφερειακό επίπεδο, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την αγροτική πολιτική ή την παιδεία. Άρα ε, σε αυτό το πλαίσιο δηλαδή σε ό,τι αφορά το διάλογο που κάνουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνουμε την υποστήριξη αυτών των ε, Δήμων και Περιφερειών. Λέγοντάς τους ότι αυτά είναι τα σημεία στα οποία θέλουμε να επιμείνουμε περισσότερο. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα τελευταίος, τελευταίο μιλήτρια έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη για το τελευταίο που είπατε. Υπάρχει ζήτηση για περισσότερη συμμετοχή στην τοπική πολιτική. Υπάρχει περιθώριο να μιλήσουμε για εφαρμογή πολιτικής, διαφάνεια, λογοδοσία των τοπικών θεσμών. Ήθελα να σχολιάσω κάποια από τα ζητήματα που αναφέρθηκαν. Πρώτον, δεν μπορούν να υπάρχουν στρατηγικές επικοινωνίες χωρίς υγιή πολιτική. Εάν ένας πρωθυπουργός ή μια πρωθυπουργός ταξιδεύει σε μια περιοχή και το μήνυμα που μεταφέρει είναι διαφορετικό, αναρνητικό για τις πρόπτικες προσχώρησης, η επίδραση θα είναι πάρα πολύ αρνητική για τις ε, στρατηγικές ε, επικοινωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης περί διεύρυνσης. Αυτό είναι το πρώτο. Θέλουμε δηλαδή συμφωνία συμμετοχή των κρατών μελών και πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η πολιτική διεύρυνση, η διαδικασία είναι αξιόπιστη και υγιής. Θα ήθελα επ' αυτού να αναφερθώ σε αυτό που είπε η δημοσιογράφος από τη Σερβία προηγουμένως. Τα μέσα, και εγώ υπερασπίζω τη συνεργασία με τα μέσα, ε, πρέπει να χαρακτηρίζονται από αντοχή, ερευνητική ε, εκπαίδευση σε θέματα έρευνα ε, και όλα αυτά. Αλλά το πραγματικό πρόβλημα σε χώρε όπω η Σερβία είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ακούν τι ειδήσει από την τηλεόραση. Και τα περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια είναι τη κυβέρνηση. Οπότε λειτουργούν ω μεγάφωνα τη κυβέρνηση. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ παρακολουθεί τη διαδικασία προσχώρηση, να εξετάζει όχι μόνο τα νομικά, τις νομικές πτυχές, αλλά και πώς πρακτικά εφαρμόζονται αυτά, ε, πώς λειτουργεί η αγορά των μέσων μαζικής ενημέρωσης πρακτικά. Διότι πολλά από αυτά συμβαίνουν παρότι υπάρχει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο, οπότε εκεί απαιτείται και η πολιτική να πηγαίνει παράλληλα με τις πρωτοβουλίες αυτές, οι οποίες είναι ξέπαινες και με τις αλλαγές που να, θα υποστηρίζει η κοινωνία των πολιτών και αλλαγές στα μέσα, αλλά χωρίς ε, να υπάρχει ένα περιβάλλον πρόσφορο για να ανθίσουν τέτοιες πρωτοβουλίες, δεν θα καταφέρουμε να επιτύχουμε αποτελέσματα. Το τελευταίο που εγώ επαναλαμβάνω διαρκώς και θα το ξαναεπαναλάβω όσον αφορά το μήνυμα που δίνουμε δεν προσπαθούμε να πουλήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια. Ο σκοπός ουσιαστικά είναι ότι τα Βαλκάνια διέρχονται μια διαδικασία μεταρρύθμισης ώστε να γίνουν υγιείς δημοκρατίες που να ανταποκρίνονται στις επιθυμίες και στις προτιμήσεις των πολιτών τους. Όλα αυτά όταν γίνονται στο πλαίσιο τη προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμφέρουν και τα Βαλκάνια και τα Δυτικά Βαλκάνια και αυτέ τι χώρε και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε σκοπό είναι να γίνουν τα, οι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων υγιεί δημοκρατίε, επίση κατάλληλε και για μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συμφέρει και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν συμφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση να πουλά μια ψευδή εικόνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήθελα να πω ως τελευταίο σχόλιο. Ευχαριστώ πολύ. Θα χρειαστεί να σας αποχαιρετήσουμε τώρα και σας ευχαριστώ όλους για την ε, συμμετοχή σας ε, στη συζήτηση. Και πάμε στο σημείο 14 της ημερησίας διάταξης. Ευχαριστώ πολύ.